Um, Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Περίμενα μέχρι να υπάρχουν αρκετά μέλη εδώ. Δεν ήθελα να αρχίσω συνεδρίαση με άδεια αίθουσα. Χάσαμε κάποια λεπτά έτσι από τις νόρες της συνεδρίασης μας. Δεν θα να περάσουμε στο σημείο της ημερησίας διάταξης, έγκριση ημερησίας διάταξης. Υπάρχουν παρατηρήσεις, διαφωνίες. Όχι, δεν βλέπω κανένα σηκώνει το χέρι του και θα ήθελα να σας πω ότι το σημείο 11 η γνωμοδότηση του κυρίου Χουντή θα εξεταστεί αύριο οπωσδήποτε. Θα με εξετάσει κατά πώ θα μπορούσαμε να το ξέρουμε σήμερα, αλλά δεν ήταν δυνατό. Θα είναι αύριο. Ο κ. Φέπε έπρεπε να το ξέρει από ό,τι κατάλαβα. Έγκριση των πρακτικών. Ωραία. Δεν βλέπω να υπάρχουν παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ανακοινώσει της Προέδρου. Έχουμε μια αίθουσα ακρόασης και σήμερα και αύριο. ΑΕΣΠ 5G2. Αν φτάσουμε λοιπόν εδώ στο αδιαχώρητο, εκεί θα πρέπει να πάνε εκείνοι που δεν έχουν βρει θέση στην αίθουσα. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είναι στο web stream οι συνεδρίες αυτές και μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση αν θέλετε και επίσης υπάρχει και μια καταγραφή βίντεο που δημοσίευσε στο Europower με 24 ώρες μετά που θα λήξει η συνεδρίαση. Αυτά για τα τυπικά. Τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να καλωσορίσω τον κύριο Eddie Wimmers Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διεθνιστικών Ερχών των Αγορών Κινητών Αξιών. Ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ κι για το θέμα αυτό. Θέλουμε να ακούσουμε τι απόψει σα και θα υπάρχει και μετά αρκετός χρόνο για ερωτήσει. Ό συνήθω. Ω συνήθω, ο Έντι θα μα κάνει μια παρουσίαση κάπου 10 λεπτά. 15 ήθελα, αλλά εγώ τον πίεσα για να μείνει στα 10 και ότι δεν θα αναφέρει θα πρέπει να αναφερθεί μετά στις ερωτήσεις. Του τον εκτένων έτυχε το λόγο. Thank you very much, Madam Chairperson. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα το ότι μου δίνει δίνετε ευκαιρία να σας ε, εξηγήσω ε, τις ε, εργασίες της Επιτροπής μας, της Επιτροπής Διεθνιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών, της ΕΡΑΚΑ. Το 2009, κυρίες και κύριοι, εργαστήκαμε πάρα πολύ σε διάφορε τομείς και θα μου επιτρέψετε να αναφέρω δύο. Ο ένας ε, τομέας ε, είναι ε, οι συστάσεις για την ρύθμιση των λογαριασμών. Εκεί συνεργαστήκαμε με την ESCB, με το Διοικητικό Συμβούλιο για την ρύθμιση, για τον έλεγχο των κινητών αξιών. Ε, υπάρχουν δύο σημεία εδώ τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχει το έγγραφο σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη προοπτική και κατόπιν υπάρχει και το θέμα που αφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Α δούμε, εν πάση περιπτώσει, τι βασικέ ε, προτεραιότητε για το 2009-2010. Νομίζω η πρώτη σημαντικότερη προτεραιότητα είναι η θεσμική μεταρρύθμιση που θα μετατρέψει την ε, ρυθμιστική, την ΕΡΑΚΑ, όπως είναι τα αρχικά, σε μια νέα μορφή θα πρέπει λοιπόν αύριο να ληφθούν οι σχετικέ αποφάσει. Το δεύτερο που έχει σημασία είναι οι οργανισμοί πιστοληπτική αξιολόγηση, όπου ξεκινήσαμε με την απόφασή μα τον Απρίλιο που λήφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χάρη των καλών σχολείων που έγιναν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίω από τον κύριο Γκοζέ, μπορέσαμε να ξεκινήσουμε τη δουλειά μα και να επιφορτιστούμε άμεσα με την εποπτεία των πιστοληπτικών οργανισμών. Στο μέλλον θα ασχοληθούμε με τους, πιστοληπτικούς, τους οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης άμεσα. Αν δούμε τώρα λιγάκι τις ε, προτεραιότητες, νομίζω ότι στη δουλειά που κάναμε σε σχέση με την κρίση υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Ε, μερικά από αυτά έχουν σχέση με την υπόθεση Λέμαν, άλλες ε, πάλι με το θέμα της απάτης ε, Μέντοφ. Ε, κατ' ουσίαν εξετάζουμε την οργάνωση των αγορών κινητών αξιών και παραγόγων και αυτό για να επιφέρουμε μεγαλύτερη διαφάνεια όπως επίσης και στην αγορά ε, μετοχών, κάτι που έχει άμεση σχέση με τη ρευστότητα. Παρεπιπτόν σας πω ότι έχουμε και αποφάσεις που θέλουμε να λάβουμε για την αγορά ομολόγων. Όλα αυτά ανησυχούν. Αυτά που ανησυχούν κυρίως είναι η λογιστική. Η δική μας, ο δικός μας οργανισμός έχει τοποθετηθεί απέναντι στο ε, Διεθνές Λογιστικό Συμβούλιο για να περιμενηθούμε τη άποψη ότι η καλή λογιστική είναι καθοριστική σημασία για τις αγορές και ε, γι' αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται και υπόψη οι αντιδράσει των αγορών. Ο φορέας μας λοιπόν δεν ασχολείται μόνο με ε, ρυθμιστικό και εποπτικό έργο. Αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία είναι ότι αναλαμβάνουμε και λειτουργικές εργασίες. Και αυτές οι λειτουργικές εργασίες επικεντρώνονται σε προγράμματα ηλεκτρονικά πληροφορικής. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε πολλούς εμπειρογνώμονες και τα προγράμματα τα ηλεκτρονικά που ε, θα εξετάσουμε σήμερα αποτελούν τη βάση δεδομένο για τους ε, οργανισμούς αξιολόγησης. Έχουμε ένα σύστημα αναφοράς και έχουμε και μία τράπεζα δεδομένων που ασχολείται με τα δεδομένα των επιχειρήσεων. Και στο τέλος θα προσθεθεί και άλλη μία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε όλα αυτά γιατί τα προγράμματα αυτά απαιτούν μεγάλα πολλά κονδύλια χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία ε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, δεν μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε αυτοχρηματοδοτηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν καταφύγαμε στους ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς για να μας ε, ε, χρηματοδοτήσουν για τη λειτουργία αυτών των συγκεκριμένων προγραμμάτων, όχι γενικότερα για τη λειτουργία της ΕΡΑΚΑ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την χρηματοδότηση των μελλοντικών μας δραστηριοτήτων. Θα ήθελα ε, να παραμείνω λίγο στο χρόνο που μου δώσατε και επιτρέψτε μου να εκφράσω κάποιες ανησυχίες που έχουμε για το μέλλον. Μία από αυτές τις ανησυχίες έχει άμεση σχέση με τη λογιστική. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν τα πηγαίνουμε και πάρα πολύ καλά στη λογιστική και έχουμε διαπιστώσει ότι τα πρότυπα πρέπει να είναι πιο αυστηρά στην Ευρώπη. Από τη στιγμή που διαμορφώνται διαφορετικά στις ΗΠΑ η ψαλίδα ανοίγει όλο και περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να αναστηθεί μια συμφωνία ανάμεσα στι δύο πλευρέ και να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα ε, το οποίο εμεί στηρίζουμε ανεπιφύλακτα είναι η εφαρμογή διεθνών προτύπων λογιστική. Θα ήθελα να αναφέρω ε, και το θέμα της ε, προστασία του επενδυτή, το οποίο βρίσκεται πολύ ψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων μα. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία θέλω να σε επισημάνω. Το πρώτο από αυτά είναι η κατανομή των προϊόντων, τα οποία εμείς αποκαλούμε προϊόντα λιανικής ε, λιανικών επενδύσεων με ε, ακρονίμιο BRIPS. Αυτά έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά είναι τα παραδοσιακά, αλλά έχουν ανασυσκευαστεί εισαγωγικά και για το λόγο αυτό διέπονται και από διαφορετικούς κανόνες. Συνεργαζόμαστε με τις δύο άλλες επιτροπές για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο καθεστώς ε, το οποίο θα αφορά όλα τα προϊόντα τα οποία οικονομικά είναι τα ίδια. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη δουλειά και νομίζω ότι ότι όλοι μας θέλουμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις δυσκολίες που υφίστανται στον τομέα αυτά. Αυτό. Όσον αφορά τώρα τα μαθήματα που εξάγαμε από τις περιπτώσεις Μέντοφ και Λίμαν, να πω το ένα έχει σχέση με τα αποθετήρια, με τις ε, παρακαταθήκες. Αυτό θα συζητηθεί αργότερα. Πρόκειται και για την οδηγία περί ε, των hedge funds, για την περίπτωση Λίμαν Εκεί ένα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι ε, μπορεί να υπάρξει κάποια βελτίωση στις, ε, στους κανονισμούς. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτό που λέω, αλλά ε, διαπιστώσαμε στην περίπτωση αυτή ότι πολλές φορές οι κινητές αξίες δεν ρυθμίζονται, η διαχείρισή τους δεν ρυθμίζεται από κανόνες. Θα ήθελα να σκεφτούμε λιγάκι και την ανάπτυξη προϊόντων, τα οποία θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα τα προϊόντα αυτά, μακροπρόθεσμα για τους επενδυτές. Ε, πρέπει να ε, προετοιμαστούμε και για τη γύρανση του πληθυσμού. Αυτό είναι σημαντικό και για την ΕΡΑΚΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών ε, Αρχών και αυτή μπορεί να συμβάλλει και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το θετικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι το ασύνηθες. Κανείς δεν έχει δει το λόγο η Αιλίν. Κοιτάξτε, δεν ήθελα εγώ να ξεκινήσω, αλλά ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα. Αυτό που με ενδιαφέρει ε, είναι αυτά που είπατε σχετικά με τα αποθετήρια και τη δουλειά που θα κάνει η Εράκα σε αυτό το θέμα. Εξ όσων γνωρίζω, στην περίπτωση Λέμαν που τη θίξατε κι εσείς, το 50% ε, είχε τοποθετηθεί ε, σε ίδια αποθετήρια και αυτό δεν επιστράφηκε ποτέ, χάθηκε. Γι' αυτό λοιπόν θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει ίσως να ζητήσετε ανεξάρτητα αποθετήρια γιατί με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει καλύτερη διασφάλιση για τον καταναλωτή και ως εκ τούτου θα υπάρχει και μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι εμείς ασχολούμεθα με τη χαρτογράφηση των διαφόρων κανόνων που διέπουν τα αποθετήρια. Κατά δεύτερον, η Κομισιόν έχει ανακοινώσει ότι θα τοποθετηθεί. Τρίτον, εγώ θεωρώ ότι στην ε, προτινόμενη οδηγία υπάρχουν κάποιοι κανόνες που αφορούν τα αποθετήρια. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτά τα αποθετήρια διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην λειτουργία των επενδυτικών ε, κεφαλαίων ε, και διότι μπορούν να βοηθήσουν στο να ελέγχει κανείς την είσοδο και την έξοδο από τα επενδυτικά κεφάλαια. Όσον αφορά τώρα την, ε, τις δραστηριότητες που μπορούν να πτύξουν τα ίδια τα αποθετήρια. Βεβαίως και αυτά αναλαμβάνουν και θα πρέπει να αναλαμβάνουν πλήρως τις ευθύνες. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν οι κινητές αξίες εναποτίθενται, παρακατε, παρακατήθενται σε δεύτερα και τρίτα μέρη. Είναι λοιπόν σημαντικότερο να περιοριζόμαστε ε, σε αυστηρούς κανόνες. Βέβαια αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Εγώ θα ήθελα, θα προτιμούσα το, τη δεύτερη περίπτωση υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί, ότι υπάρχει αυστηρή επιτήρηση και δεύτερον να υπάρχει επιπρόσθετα και αυτό που αποκαλούμε κανόνες επίπεδου 3 οι οποίοι ισχύουν όσον αφορά την ε, λειτουργία των ταμείων. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι για να διασφαλιστούν οι κινητέ αξίες ε, στα αποθετήρια σε όλο τον κόσμο, αυτό σημαίνει πολύ μεγάλο κίνδυνο. Οι κίνδυνοι πρέπει να ασφαλίζονται, αυτό κοστίζει και δεν είναι και απαραίτητα προ όφελο του επενδυτή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντως ε, η μεταρρύθμιση της εποπτείας ε, της δημοσιονομικής στην Ευρώπη ήταν κάτι αναμενόμενο ε, όχι μόνο λόγω της δημοσιονομικής κρίσης αλλά επειδή υπέρχει λόγος και έχει καταδείξει η Ευρώπη ότι είναι διατεθειμένη να αναλάβει τις ευθύνες ό,τι αφορά την εποπτεία του δημοσιονομικού συστήματος. Έλαβε τώρα συγκεκριμένη μου μορφή αυτό, επιβεβαιώθηκε και στο Πίτσμπεργκ εφόσον ελήφθη η απόφαση να ε, ενδυναμωθεί, να ενισχυθεί αυτή η εποπτεία. Η δημοσιονομική κρίση που μας έπληξε το 2008 ε, εξέπληξε όχι μόνο τους εθνικούς αλλά και τους ευρωπαίους επόπτες. Μας έδωσε τη δυνατότητα έτσι να καταλάβουμε τα ελλείμματα που είχαμε ε, σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική της δημοσιονομικής υποπτίας. Τι έγινε λοιπόν ενάντια της κρίσης στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, στα δημοσιονομικά όργανα έλαβαν κατακριματισμένες αποφάσεις, ε, ήταν έκδηλη η έλλειψη συντονισμού. Η δική σας ε, οργάνωση είναι συμβουλευτική κύριε Πρόεδρε προς το παρόν και δεν είχε προφανώς τις επαρκείς αρμοδιότητες για να συνεισφέρει περισσότερο στην ε, εξέβρεση λύσεων. Παρά την εμπειρογνωμοσύνη την οποία έχετε πολλάκις αποδείξει ότι κατέχετε Όλα τα θεσμικά όργανα λοιπόν θα πρέπει να συνεισφέρουν ε, με δεσμευτικό τρόπο, δηλαδή η άποψή τους να είναι δεσμευτική, γιατί πολύ καλή είναι η εμπειρογνωμοσύνη, πολύ καλές είναι οι συμβουλές, αλλά η δεσμευτική ε, ευθύνη που έχει κάποιος όταν αναλαμβάνεται είναι πολύ πιο ε, σημαντική. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι απλό, Πρόεδρε, κατόπιν τούτων. Μπορείτε να μας πείτε σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας Μπορείτε να μας πείτε λέγω περισσότερα στοιχεία για το νέο όργανο που θα αντικαταστήσει τη δική σας Επιτροπή για την εποπτεία των δημοσιονομικών αγορών και οι νέες αρμοδιότητες που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρείτε ότι θα είναι επαρκής για τη διασφάλιση μιας κάποιας σταθερότητας των δημοσιονομικών ε, αγορών των οποίων η αστάθεια έπληξε όπως ξέρουμε όλοι με οξύ τρόπο την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς να απαντήσω ή στην αγγλική ή στη γαλλική. Στη γαλλική θα προσπαθήσω παρόλο που δεν είμαι γαλλόφωνος. Για την αυριανή συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών είναι πολύ σημαντική η πρόοδος που έχει γίνει. Δηλαδή πρώτη φορά ένα θεσμικό όργανο ε, θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά για την εποπτεία των δημοσιονομικών ε, των χρηματαγορών. Είναι ένα πρώτο βήμα βεβαίως. Και προφανώ όχι το τελευταίο. Είμαστε στην αρχή ακόμα τη διαδικασία. Ε, είναι η προσέγγιση Ντελαροζιέρ, η οποία είναι συνετή, μετριοπαθή και νομίζω ότι στα πλαίσια αυτά έχουμε πολύ σημαντικά περιθώρια προόδου. Πολύ σωστά τώρα θέσατε έμφαση ε, το δεσμευτικό κομμάτι των προτάσεων αυτών. Νομοθετικά δεσμευτικό. Όντως, αυτό που μας έλειπε μέχρι τώρα ήταν η δυνατότητα να επιβάλλουμε ορισμένες αποφάσεις. Από τον Οκτώβριο του 2008 Έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε αποφάσει στον τομέα αυτό με ειδική πλειοψηφία. Και το κάναμε ήδη από την πρώτη μα ε, συνάντηση, από την πρώτη μα συνεδρίαση. Η θεσμική αυτή αλλαγή, δηλαδή η δική πλειοψηφία στη θέση της ομοφωνίας, είναι ήδη μία πρόοδος για την επιβολή κάποιων αποφάσεων. Τώρα θα πρέπει να περάσουμε σε μεγαλύτερη ταχύτητα. Μεγαλύτερη ταχύτητα που προβλέπεται από την πρόταση που θα συζητηθεί αύριο στο Συμβουλίο των Υπουργών. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε εκτό αν το θέλετε. Μπορώ να μπω σε λεπτομέρειε στι διαφορετικέ πτυχέ των προτάσεων, αλλά εγώ τα εξή δύο θα ήθελα να τονίσω. Πρώτον, να υπάρχουν κανόνε βεβαίω τεχνική φύσεω Βεβαίως όχι πολιτικής φύσεως, είναι προφανές αυτό, τεχνικής λοιπόν φύσεως, αλλά νομοθετικά, νομικά δεσμευτικές. Και νομίζω ότι για αυτό το θέμα είμαστε στον καλό δρόμο. Έχουμε κάποιες ε, επιφυλάξεις, αλλά μπορέσουμε να τις συζητήσουμε αργότερα. Και κατόπιν, δεύτερο, να ελέγχουμε την πραγματική και αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των κανόνων. Μέχρι σήμερα έχουμε πολλού κανόνε σε όλου του τομεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι εφαρμόζονται πάντα με τον επαρκή και κατάλληλο τρόπο. Και έτσι μπορεί να παρέμβει αυτή η νέα υπηρεσία για να εντοπίσει τα κενά με μια διαδικασία βεβαίω που θα σέβεται τα δικαιώματα όλων των ενδιαφερομένων φορέων, αλλά τελικά να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει στι εθνικέ αρχέ, αγαπητοί φίλοι, δεν κάνατε αυτό που έπρεπε να κάνετε, να το κάνετε αν δεν το κάνετε, και βεβαίω αυτό είναι πολύ επίμαχο ε, σημείο, αν δεν το κάνετε, εγώ, εγώ η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα υποκαταστήσω την Εθνική Νομοθεσία. Βεβαίω ξέρω ότι είναι επίμαχο το ζήτημα αυτό. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν αύριο στο Συμβούλιο τα κράτη-μέλη. Ό,τι όμω και να γίνει, πιστεύω ότι η πρόοδο είναι σημαντική. Έφεξης, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο περιθώριο παρέμβασης θα πρέπει να οικοδομήσουμε τη νέα αυτή αρχή, όπως αναφέρεται, με προσωπικό, με μέσα να την προκοδοτήσουμε, να δούμε τις πηγές χρηματοδότησης, αλλά για αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα, σε αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητήσει τον ε, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Βάιμαρσε. Ε, θαυμάσια είναι, είναι αυτές οι διαφάνειες που μας δείξατε και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον εσείς στηρίζετε ε, την, το κέρδος ε, κατά πόσον όσον αφορά το κέρδος αναμετοχή αν θα πρέπει να υπολογίζεται με την πραγματική αξία ή ε, με την ερμηνεία ορισμένων. Ε, το διάβασα κάπου αυτό και δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει το πρέπει το αναφέρατε, ε, ίσως αξίζει τον κόπο να το εξετάσουμε και οτιδήποτε πρέπει να κάνουμε για να υπάρχει μεγαλύτερη κατανοηστή ε, και μεγαλύτερη διαφάνεια. Όσον αφορά τη γύρανση, χαίρομαι που τα αναφέρετε όλα αυτά. Διάβασα ότι το 2010 το 75% ε, του εισοδήματος στην Ευρώπη θα είναι για άτομα πάνω από την ηλικία των 50 ετών. Ε, αυτό όμως σημαίνει μια μεγάλη εξέλιξη και γι' αυτό θα ήθελα να γνωρίζω πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους ε, στα γυρατιά τους και πώς να ε, πείσουμε τους νέους να αποταμιεύουν. Γιατί αυτοί που αποταμιεύουν δεν θα τους φτάσουν όταν θα είναι πια ηλικιωμένοι, γιατί είναι μεγαλύτερο το προσδόκιμο ζωής. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και ευχαριστώ που αναφέρατε και τη γύρανση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο διότι με ενδιαφέρει πολύ. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για το μέλλον. Ένα μακροοικονομικό ερώτημα. Θα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε νέα μέσα τα οποία να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων. Δηλαδή, να ξέρουν ότι θα αποδώσει η σύνταξή τους, όποια μορφή και αν έχει, κρατική, ιδιωτική ή οτιδήποτε άλλο. Και έτσι το συνδέω αυτό με το ΠΡΕΠΣ. Έχουμε μια σειρά προϊόντων και συνταξιδοτικών, περισσότερο ενδεχομένω ε, ε, στις Βρετανικές νήσους από ότι στην υπηρετική Ευρώπη, που δεν προσφέρονται υπό τις ίδιες συνθήκες σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες, τις συμβουλές, την δημοσίευση των αμοιβών κτλ. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ισότιμη βάση, να διασφαλίσουμε ισότιμη βάση. Ούτω ώστε οι επενδυτέ, διότι και οι μελλοντικοί συνταξιοδο... συνταξιοδοτούμενοι είναι επενδυτέ. Να γνωρίζουν πού πηγαίνουν. Το θέμα αυτό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν θέλω να λάβω θέση. Δεν θέλω να τοποθετηθώ. Και το βασικό που θέλω να πω στους εμπειρογνώμονες είναι παρακαλώ να βρείτε μια λύση κύριοι και κυρίες εμπειρογνώμονες που να γίνει αποδεκτή από όλους. Να είναι συνενετική. Να μην την ασπαστεί ένα κομμάτι του κόσμου και να την απορρίψει άλλο. Διότι αλλιώς θα προσκρούσουμε στα ίδια προβλήματα πάλι. Ευχαριστώ. Ε, Κύριε ε, θίξατε αυτό το θέμα της ε, λογιστικής, προτύπων για τη λογιστική. Εγώ δεν θέλω να εμβαθύνω σε αυτό, να σας αναφέρω όμως μόνο ένα παράδειγμα. Η Deutsche Bank, η γερμανική αυτή τράπεζα, έχει 1,83 ισολογισμός, ε, ισολογισμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Και σύμφωνα όμως με αμερικανικά πρότυπα, 950 δις αντί για 1,83. Δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο, μια τεράστια διαφορά.

Και αυτό το άκουσα πριν από τρία χρόνια από τον κύριο Μακρύβη και από τον Γενικό Διευθυντή του τότε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο ε, κάπου να συναντηθούμε στα πρότυπα ενώ με τους Αμερικανούς ε, και να ξεπεραστεί αυτό το χάσμα. Σήμερα όμως ε, έχω καταλήξει περισσότερο στο ότι αποκλίνουμε. Δεν συγκλίνουμε, αποκλίνουμε. Γι' αυτό λοιπόν ξεχάστε το fair value, τις δίκες αξίες ή όχι, αλλά ε, σωστά ε, λειτουργεί το σύστημα και σε ποιον είμαστε υπόλογοι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν είμαστε υπόλογοι σε κανένα. Είμαστε ένα είδος ε, υπτάμενης οντότητας και δεν αποδίδουμε λογαριασμό πουθενά. Κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά θέματα επιτάπητος, δεν γίνεται αλλιώς, είναι μεγάλη πίεση και πρέπει να υπάρξει σκληρή δουλειά. Και αυτό οδηγεί στο ότι εν μέρη προσπαθούμε να απαντήσουμε σε θέματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με άλλα θέματα τα οποία ε, δεν μπορούμε όμως να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Έχω κατά νου ε, τα αποθετήρια και depository passport για IFM και παράλληλα έχουμε και το θέμα των deposit usage. Φτάνουμε λοιπόν ίσως σε μία λογική όπου πλέον ε, τα πράγματα αυτά δεν συνδέονται, τουλάχιστον σίγουρα όχι όσον αφορά τη χρήση, usage. Και το τελευταίο που θέλω να πω, ε, ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση. Αυτή η οδηγία περί προοπτικής έχει νόημα να εξεταστεί τώρα όταν ξέρουμε ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε το PREPS και το PREPS ε, θα είναι κατ' ουσίαν η προσπάθεια προσπάθεια να αναπτύξουμε καινούργια προϊόντα. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε το τελευταίο γιατί είναι το πιο απλό. Λέτε ότι το πρίψει είναι ένα καλό παράδειγμα. Η φυστάμενη πρόταση για τα πρίψη δεν πάει τόσο μακριά όσο στην οδηγία α, για το perspective τις προοπτικές. Σε ορισμένα συγκεκριμένα σημεία θέλουμε ίδια μεταχείριση για τα συγκρίσιμα προϊόντα. Η συγκρίσιμη μεταχείριση για τα ίδια προϊόντα. Αυτό στην οδηγία Prospective περιορίζεται μόνο στα short perspective, στην βραχυπρόθεσμη προοπτική. Δεν υπάρχουν δηλαδή, δεν υπάρχει το πλήρες φάσμα των προοπτικών για όλα τα προϊόντα. Πέραν τούτου, ορισμένοι κανόνες που αφορούν τα MIFID μπορεί να είναι χρήσιμες και για άλλα προϊόντα. Οι πρίψη λοιπόν και οι προοπτικές έχουν κάποιες άλλες επικαλύψεις, έχουν κάποια κοινά σημεία, αλλά όχι βεβαίως εντελώς, δεν είναι το ίδιο. Για τα deposits τα... Ε, ε, συμφωνώ ότι υπάρχει φαινόμενο μετάγγισης spillover effect όπως το λέμε είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά, πιστεύω ότι είναι αναπόφευκτο και εξαρτάται και από εσά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή ε, να ε, νομοθετήσετε ούτω ώστε να υπάρχει αρμονική συνύπαρξη των διαφόρων. Διότι προς το παρόν δεν υπάρχει. Και αυτό είναι κομμάτι της συζήτηση που έχουμε και είχαμε και κατά το παρελθόν. Τώρα, για το ISB. Η συζήτηση αυτή για την απόκληση ή τη σύγκληση. δεν είναι ο μόνος τομέας στον οποίο υπάρχει αυτό. Το βλέπουμε και στα λογιστικά, το βλέπουμε και στα παράγωγα, το βλέπουμε και στα hedge funds. Υπήρχε το Caesar πριν από κάποια χρόνια, Όπως συζητούσαμε ε, ενεργά με τους Αμερικανούς την αμοιβαία αναγνώριση. Όμως με την κρίση μπήκε τέρμα σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ήμουν την περασμένη εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη, στη Ουάσιγκτον και είπα ότι είμαστε ακόμα αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε την αμοιβαία αναγνώριση, ότι αυτό είναι το μέλλον. Και από του Αμερικανού το ίδιο κατάλαβα, ότι του ενδιαφέρει να το εφαρμόσουν παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά υπάρχει κρίση, όπω είπα πριν, αφενό που πλήττει περισσότερο τι δομέ, τα θεμέλια τη οικονομία μα από ό,τι πέρσι, φέτο και δύο, αφετέρου, η ΕΠΑ έχουν να κάνουν μια θεσμική μεταρρύθμιση που δεν ξέρουμε ακόμα πού θα φτάσει και προς τα πού θα πάει. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συζητήσουμε με τους Αμερικανούς. Για το ISB δεν είπα τίποτα. Όντως, όντως, ε, συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι θα πρέπει η διακυβέρνηση των ISB να επανεξεταστεί το πραγματικό θέμα αυτό είναι. Η διαχείριση αυτή, η αυτοδιακυβέρνηση του τομέα είναι ισορροπημένη. Στην Επιτροπή Σίζαρ είχαμε πει ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες μεταλλαγές τόσο ώστε να οδηγηθούμε σε μια πραγματική ελεγκτική επιτροπή, επιτροπή εποπτείας. Εγκαταλείφθηκε αυτή η ιδέα προς το παρόν. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να ξανατεθεί. Εξ αρχής.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 pero cuando se llega a poner esto negro sobre blanco, como decía un poeta español, de pasar de las musas al teatro, las, las divergencias afloran. El gran problema es las decisiones dirigidas por la autoridad bancaria o la autoridad de supervisión de mercado. Θα προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε μέσα από άλλη καμπίνα. Εντάξει, λοιπόν, ε, θα ήθελα, γιατί δυστυχώς από... έχει μεγάλο μικροφωνισμό. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι όταν υπάρχει ένα εθνικό όργανο το οποίο δεν λειτουργεί σωστά, ε, δεν θα πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικοί κανονισμοί. Στην περίπτωση αυτή, μήπως ε, θα πρέπει ο οργανισμός αυτός να καταφύγει ε, σε ιδιώτες σε έναν τομέα ο οποίος μέχρι τώρα δεν καλύπτεται από κανονισμούς και πρότυπα. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, τι ακριβώς πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μην υπάρχει ε, αυτό το αποστηρωμένο περιβάλλον. Φαντάζομαι ότι και εσείς ε, δεν θα μπορείτε να πείτε πολλά πράγματα από αυτό αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να γνωρίζω τη δική σας την εμπειρία, τι ακριβώς πιστεύετε κυρίως ε, στις ε, ακίνητες αξίες, γιατί αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην Ισπανία. Είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες εκπλήξεις, κυρίως όσον αφορά την φερεγγιότητα ορισμένων επιχειρήσεων. Όσον αφορά το θέμα του δημοκρατικού υπολογίου που δικαίως το αναφέρατε, Υπάρχουν κάποιες ε, προβλέψεις στον προτινόμενο κανονισμό που αφορούν αυτό το θέμα της δυνατότητας ε, του να είναι υπόλογη ένα τμήμα της ε, προσπάθειας αυτής είναι η σημερινή ακρόαση. Και στο μέλλον θα πρέπει όχι μόνο να συνεχιστεί, αλλά και να ενδυναμωθεί. Τούτου λεχθέντος θεωρώ ότι όλοι μας οι συνάδελφοι στις, ε, στα τρία θεσμικά όργανα πιστεύουν ότι θα πρέπει νομικά να μην ε, προδώσουν την ανεξαρτησία τους. Η ανεξαρτησία βασίζεται σε εθνική, στην εθνική ε, δικαιοσύνη και θα ήταν πολύ δύσκολο να υπάρχει παρέμβαση παραδείγματος χάρη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τρόπο τον οποίο να ασκούν τα καθήκοντά τους και γι' αυτό εξακολουθούμε να είμαστε αντίθετοι στο να παρέμβει η Κομισιόν στους τροποποιήσεις των τεχνικών προτύπων. Γιατί ξέρετε, τα τεχνικά πρότυπα θα βασίζονται στα λογιστικά πρότυπα και η Κομισιόν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει. Και αυτό βέβαια είναι μια παρέμβαση στην ανεξάρτητη θέση και στον ανεξάρτητο ρόλο των αρχών και των εθνικών ε, εποπτών. Απ' την άλλη μεριά ρωτήσατε κύριε Γκαρθία Μακάλο για την ρήτα διασφάλισης σε περίπτωση διαμεσολάβησης. Σύγκριση δηλαδή συμφερόντων μεταξύ διαφόρων αρμοδίων αρχών. Βλέπω ότι η προτινόμενη πρόταση λέει ότι στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει μια απόφαση από ένα πάνελ που θα αποταθεί στους εθνικούς επόπτες. Ένα αυτό. Θέλουμε να έχουμε μερίτρα διασφάλιση για φορολογικές ευθύνες γενικά, αλλά είπαμε ότι αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να εξεταστεί βάση του άρθρου 23, όχι να αφορά τη διαμεσολάβηση, γιατί από ό,τι κατάλαβα για τη διαμεσολάβηση, η απόφαση ε, του Συμβουλίου Εποπτείας, εάν δεν εφαρμοστεί, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Και ε, αυτό σχετίζεται βέβαια με μια νομική απόφαση. Και το μόνο που μπορεί να γίνει θα είναι να υπάρχει παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και στην περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή θα μπορεί να προσφύγει στα εθνικά δικαστήρια για να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Απόφαση. Θα δούμε όμως τι θα αποφάσει. τελικά η πολιτική. No. That's the, not, nothing about accounting because you say solvency. Κοιτάξτε, αναφερθήκατε στα καθόφλια ρευστότητα. Ε, ε δεν ξέρω ακριβώ τι εννοείται, αλλά αυτό είναι θέμα των τραπεζικών αρχών και γι' αυτό έχω τη δικαιολογία να μην σα απαντήσω. Πρόεδρο, ωραία. Κύριο Πούλμαν. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ που απαντάτε εδώ στις ερωτήσεις μας. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο για την συζήτηση που είχατε μόλις τώρα με τον συνάδελφο Γκαρσία Μαγκάλο όσον αφορά τα τεχνικά πρότυπα και την εξέτασή τους. με τον ε, δημοκρατικό έλεγχο θα μπορούσε να φανταστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές δυνατότητες ε, προετοιμασίε αυτών των τεχνικών πρότυπων με επιτροπέ εθνικών υπερογνωμένων με ανάμειξη κομισιών κλπ. Αυτό που δεν μπορούμε να φανταστούν είναι ότι τεχνικά πρότυπα θα ε, υιοθετούνται χωρί να δράσει πλήρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ασκήσει το δικαίωμά του να ελέγξει το τελικό αποτέλεσμα. Και να παρέμβει μονάχα όταν έχει ε, υπάρξει αρνητικό αποτέλεσμα για την οικονομία. Αλλά αυτό το θέμα θεσμική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ίσω ένα άλλο σχόλιο από πλευρά σα για το θέμα αυτό, γιατί αυτό νομίζω ήταν και ησυχία του κυρίου Γκαρσία Μαργκάλιο. Και κάτι άλλο όσον αφορά τα προϊόντα στα οποία αναφερθήκατε, δεν θα σας παρακαλέσω να το διευκρινίσετε λιγάκι. Πώς η πρότασή σας για περισσότερη διαφάνεια στην αγορά αυτών των προϊόντων θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Θα ακολουθήσουμε μόνο τα πιο τυποποιημένα προϊόντα και τι θα γίνει με τα μη τυποποιημένα προϊόντα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Πώς θα συμμετάχουμε εκεί στον κίνδυνο. Για την πρώτη σας παρατήρηση έχω να πω ότι αυτή είναι πολιτική και ω πρόεδρο μια επιτροπή που είναι τμήμα ε, Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου δεν θα τοποθετηθώ. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσετε εσεί με του συναδέλφου από τα άλλα δύο πολιτικά σώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, ότι αυτό δεν είναι θέμα δικό μου να απαντήσω, αλλά η άλλη ερώτηση. Ναι, συζητάμε για τεχνικά πρότυπα. Και το θέμα που θα τεθεί θα είναι τι είναι τεχνικό πρότυπο. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. στο τραπεζικό σύστημα έχουμε κάποιες προδιαγραφές για ε, παρουσίαση των αποτελεσμάτων στις ευρωπαϊκές αρχές, πράγμα που γίνεται με πολύ διαφορετικές μεθόδους. Δηλαδή, υπάρχει για κάθε περίπτωση ένα ορισμός Και οι ορισμοί αυτοί είναι διαφορετικοί. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τις αναγνωρίσουμε τους ορισμούς αυτούς κατά το δυνατόν. Και το θέμα που τίθεται είναι, εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο θα ορίσετε. Θα χρειαστείτε κάθε χρόνο δύο χρόνια να το πούμε έτσι για να το καταφέρετε. Ε, το θέμα του ελέγχου είναι θέμα πολιτικού ελέγχου και όχι ε, πρακτικού ή τεχνικού και θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι πολιτικοί στόχοι, ποιε είναι οι πολιτικέ προοπτικέ. Εκεί μπορεί να γίνει διάλογο. Και αυτό το διάλογο θα το ανέχουμε με όποιο ενδιαφέρεται. Αν θέλετε να με καλέσετε μεθαύριο, δηλαδή, αν είσαι τώρα εδώ. Αναμονούνται τι. Items are... Ναι. Τι κάνετε με τα παράγωγα προϊόντα. Ποια είναι τα συγκεκριμένα σημεία που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις εκθέσεις αυτές που παρουσιάζονται. Αλλά το θέμα είναι, υπάρχει παρουσίαση, υπάρχει, πώς ε, διαδίδονται αυτές οι εκθέσεις. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι. Και μια που ξεκίνησα για τα παράγωγα, να σας πω και κάτι άλλο. Πριν από μερικού μήνε δημοσίευσε η Κομισιόν ένα έγγραφο, τον Οκτώβριο νομίζω, το οποίο υποστηρίζουμε πολύ, γιατί κινείται νομίζω προ σωστή κατεύθυνση και θα θέλουμε πραγματικά κάτι να γίνει στον τομέα. Υπάρχουν διάφορα σημαντικά θέματα εκεί. Το πρώτο και κυριότερο είναι πώς μπορούμε να μειώσουμε το κίνδυνο στην αγορά παραγόγων προϊόντων. Δεν μιλάμε εδώ για δις και εκατοντάδες ε, ε, δις, αλλά για τρεις εκατομμύρια και πολλά, όχι ένα και δύο. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε με ό,τι κάνουμε να μην καταστρέψουμε την κοινωνία μα Υπάρχει κίνδυνος. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μέχρι στιγμής βρήκαμε διάφορους μηχανισμούς που ακολουθούν την ίδια γραμμή λίγο πολύ. Δηλαδή προσπαθούν να απλουστεύσουν την κατάσταση και το κάνουμε αυτό στο CCP, Central Counterparts. Δημιουργήθηκε αυτό το Central counterparties και για μετοχές και για παράγωγα και αυτό μειώνει τον κίνδυνο. Και έτσι μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ε, οι αγορές αυτές λειτουργούν επαρκώς, βάσιμα και με τρόπο με τον οποίο δεν οδηγούμεθα σε προβλήματα και θέλουμε να έχουμε μια σειρά συστημάτων που χρειάζεται χρειαζόμαστε για να μπορούμε να στηρίξουμε αυτά τα central counterparties, τα CCPs. Τώρα, τυποποίηση. Δεν μπορεί κανένα να αντισταθμίσει εκείνα τα συμβόλαια που είναι τυποποιημένα. Δεν μπορεί να κάνει κανένα τίποτα για να αντισταθμίσει το προϊόν Α με το προϊόν Β που είναι τελείως διαφορετικά. Θα πρέπει τα προϊόντα αυτά να είναι συγκρίσιμα για να μπορούν να αντισταθμίσουν το ένα το, άλλο. Τώρα πώς θα είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει αυτή η τυποποίηση. Οι αγορές δεν θα χαρούν ιδιαίτερα βέβαια. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη απόδοση από τα μη τυποποιημένα προϊόντα. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι υπάρχει τυποποίηση αυτή και θα το κάνουμε με διαφορετικούς τρόπους. Και το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Στη ΣΥΠΑ εξετάζουν αυτό να γίνεται με απόφαση κυβέρνηση. Μία προσέγγιση είναι αυτή. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Παραδείγματο χάρη, στα ενία ονόματα, αν έχει κανένα συνδέσει για κάποια ονομασία, θα πούμε ότι αυτό είναι η τυποποιημένη ε, περίπτωση. Λίγο πολύ τέλο πάντων. Αυτό θα μπορεί να γίνεται μέσω αυτών των τεχνικών ε, προτύπων, το οποίο συζητήσαμε. Αλλά εκτό αυτού, και βλέπω ότι η προτάσει τη Κομισιόν Κοινού προ μια διαφορετική κατεύθυνση, να επιβάλλουμε απαιτήσει κεφαλουχικού τύπου για μη τυποποιημένα προϊόντα. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να περάσει από το CCP θα πρέπει να είναι πιο ακριβό, να πληρώνεται περισσότερο. Και οι δύο προσεγγίσεις αυτές δεν είναι ασύμβατες μεταξύ τους. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Τις ερωτήσεις του κύριου Στόλογιάν και μετά εγώ κάποιος θα απαντήσουμε σε όλες μαζί. Κοιτάξτε, ε, πρέπει να ομολογήσω ότι έχω κάποιες ε, δυσκολίες στο να κατανοήσω τα αίτια αυτής της κρίσης. Και θα ήθελα να υποβάλω μια πολύ απλή ερώτηση. Ποια είναι τα επιχειρήματα, τα κίνητρα που οδήγησαν στο ότι πολλές ε, δραστηριότητες με τοξικά απόβλητα όπως ε, αναφέρονται δεν εμφανίστηκαν στους ε, ισολογισμούς των οικονομικών οργανισμών και έγινε αποδεκτό να κρατούνται αυτά τα απόβλητα εκτός των συλλογισμών και των τραπεζών και άλλων οργανισμών. Κοιτάξτε, ε, και εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση σε σχέση με αυτά που κάνατε, τα CCPs, όπως είπατε, τα Central Counterparties. Ε, υπάρχουν οι διατάξεις ε, περί φερεγγιότητας ή ικανότητας ε, πληρωμών. Ε, και οι εγγύησει. Αυτά όμως από μόνα τους δεν, γίνονται, δεν θα μπορούσαν να μετραπούν συστημικά στην επόμενη κρίση. Γιατί πρέπει να σας πω ότι και εγώ ίδια ανησυχώ λιγάκι από αυτού. Και επίσης διαρωτώ με κατά πόσον θα θέλατε να πείτε ε, κάποια περισσότερα λόγια για τα περίφημα dark pool κατά πόσον αυτά ασκούν μεγάλη επιρροή στην αγορά ή μήπως ε, θα πρέπει όλα να είναι μονίμως και πάντα ορατά. Κατόπιν, όσον αφορά την αναδιάρθρωση των προϊόντων, πιστεύετε εσείς ε, ότι μερικές φορές ε, λαμβάνει χώρα πολύ μεγάλη μορφή αναδιάρθρωσης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο κατά την άποψή μου ε, θεωρείτε ότι εσείς το έχετε, μάλλον εσείς πιστεύετε ότι έχετε λύσει το πρόβλημα κυρίως όσον αφορά τη σύγκρουση των συμφερόντων. Ε, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα εξετάσω τις ερωτήσεις σας ε, κατά σειρά. Πρώτον, γιατί αυτά τα τοξικά κεφάλαια εξακολουθούν να υπάρχουν στους ισολογισμούς των ε, τραπεζών. Ε, πρώτον, γιατί αγόρασαν οι τράπεζες αυτά τα προϊόντα και εφόσον το έκαναν γιατί τα κράτησαν. Το πρώτο που παίζει ρόλο είναι ότι αυτά τα τοξικά προϊόντα ε, δισέδισαν ε, στις, ε, στους συλλογισμούς των τραπεζών γιατί είχαν καλύτερη απόδοση από ομόλογα και άλλα προϊόντα. Άρα δηλαδή ήταν θέμα καθαρά απόδοσης. δεύτερον, οι τράπεζες, σωστά ή λάθος, εσείς θα το κρίνετε, βασίστηκαν στην αξιολόγηση και όπως ξέρετε αυτά τα προϊόντα, πολλά από αυτά έχουν αξιολόγηση 3α όπως είναι και τα κρατικά ομόλογα. Ε, για συστήματα τέτοια με 3α δεν υπάρχει σχεδόν καμία προϋπόθεση καθόλου κεφαλαϊκής επάρκειας. Άρα δηλαδή το σύστημα είναι εκείνο το οποίο οδήγησε σε αυτή την πολύ θλιβερή κατάσταση όπου τα τοξικά προϊόντα μπήκανε στους ισολογισμούς και από τη στιγμή που άρχισαν να ε, πολλαπλασιάζονται και να διωγγώνονται κατέρευσε το σύστημα. Ένα μεγάλο μέρος ευθύνης φέρουν οι οργανισμοί αξιολόγησης και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί τουλάχιστον σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τέτοιου είδους ε, περιπτώσεις. Κατόπιν, πιο δύσκολο είναι το ερώτημα κατά πόσον τα CCPs, ε, τα counterparts, ε, central counterparts, ε, είναι η λύση του μέλλοντος. Εγώ πιστεύω πως ναι, γιατί είναι πολύ ορατά. Βεβαίως, ο κίνδυνος σωρεύεται στην αγορά και ο κίνδυνος αυτός πλέον δεν συγκεντρώνεται στα CCPs. Είναι μια σώρευση, θα πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός στη διαχείριση κινδύνου όσον αφορά τα CCPs. Και αν τελικά συμβεί κάτι σε ένα από αυτά τα CCPs, αυτό είναι ένα θέμα όπου πράγματι ε, προκύπτει ε, συστημικός κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, αλλά ίσως ε, κάποια στιγμή ελπίζω ε, κάποιος ε, θα μπορέσει να παρουσιάσει συστήματα διαχείρισης κινδύνων που θα είναι πιο τελειοποιημένα και καλύτερα από αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς. Αν δεν αισθάνεστε και πολύ άνετα, συμφώνα μαζί σας, αλλά δεν έχω να σας δώσω μια καλύτερη απάντηση όσον αφορά τα περίφημα dark pools. Κοιτάξτε, η συζήτηση είναι πολύ περίεργη. Δημιουργεί σύγχυση, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, ούτε τον όγκο του, ούτε ξέρουμε γιατί είναι σκοτεινά. Δεν ξέρουμε γιατί οι άνθρωποι μετακινούνται στο ένα και μετά στο άλλο άκρο της αγοράς. Όπως λέτε, ε, θα πρέπει ε, να ληφθεί υπόψη ε, κατά πόσο είναι δυνατόν να εκτελούνται παραγγελίες ή εντολές χωρίς να επηρεάζεται η αγορά. Μια μεγάλη εντολή βλέπουμε ότι κατακαιρματίζεται πολλές φορές σε μικρότερες. Δηλαδή αν κάποια μεγάλη ε, σε μικρότερες εντολές αυτό δεν επηρεάζει την αγορά. Υπάρχουν όμως πολλά πράγματα που δεν είναι απόλυτα σαφή και εμείς ε, το θέμα αυτό το μελετάμε. Ελπίζουμε σύντομα να καταθέσουμε γνωμοδότηση. Δεν λέω βέβαια ότι πρέπει να ρυθμίσουμε τα περίφημα dark pool Απλά λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνουμε και πολύ καλά. Πρέπει να έχουμε καλύτερα στοιχεία για να δούμε τι ακριβώς διαδραματίστηκε κατά δεύτερον για να γνωρίζουμε ακριβώς και το διακύβευμα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σας ομολογήσω ότι δεν έχω να σας δώσω τη σωστή απάντηση. Η τελευταία σας ερώτηση κυρία Πρόεδρε αφορά στην αναδιάρθρωση καλύτερα αναδιάρθρωση παρά αποπληρωμή του χρέους. Κοιτάξτε, στον τομέα των ε, επενδυτικών κεφαλαίων, εμένα μου αρέσει καλύτερα η αναδιάρθρωση και οι συγχωνεύσεις. Γιατί στην Ευρώπη έχουμε πάρα πολλά μικρά επενδυτικά κεφάλαια. Παρεπιπτόντως, η USITS 4 επιτρέπει ε, πιο εύκολα την συγχώνευση των ε, επενδυτικών κεφαλαίων κατά πόσον εκεί θα υπάρχουν ε, προμήθειες ή όχι, δεν το ξέρω, αλλά τα επενδυτικά κεφάλαια έτσι κι αλλιώς πάντα σχετίζονται με προμήθειες. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε που ενδεχομένως δεν έχουμε σκεφτεί εμείς. Πολλά δεν είχαμε τη δυνατότητα να αναφέρουμε. τα short selling rules, ή κανόνες της α, ε, α, ε, βραχίας πώλησης. Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση τους, αλλά προκαλούν σύγχυση. Πάντως και για την αποκάλυψη πληροφοριών και για την ελεύθερη χρήση ε, προσπαθούμε να ρυθμίσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν οι ομολογίες ε, διαθέσιμες, δεν μπορείτε να πουλήσετε ένα προϊόν. Με άλλα λόγια, αέρα. Είναι όμως μεγάλο ζήτημα και αν το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται να ακούσει τι κάνουμε από αυτού, με τα χαρά να σας τα πω. Βεβαίως, βεβαίως, με το πλήρωμα του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ εκ νέου και σας ε, περιμένουμε την επόμενη φορά με μεγάλη χαρά. Ο λίγων λεπτών διάλειμμα για να προετοιμαστούμε για το επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Η έκθεση της κυρίας Άλβαρεθ.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 Σα Σας ευχαριστώ. Όπως είπα, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Έχουμε ένα σχέδιο εκθέσεως από την εισηγήτρια Μαγδαληνή Άλβαρεθ. Σας είδα κύριε Άλβαρεθ, αλλά θα παρακαλούσα όσοι θέλουν να συζητήσουν ή να τυρβάσουν επί άλλων θεμάτων παρακαλώ να αποχωρήσουν. Παρακαλώ λίγη ησυχία συνάδελφοι. Παρακαλώ. Η κυρία Άλβαρεθ. Ευχαριστώ. Στην προηγούμενη μου παρέμβαση στην ανταλλαγή απόψεων, εξέφρασα τη ρητή μου άποψη για την διοικητική συνεργασία στον φορολογικό τομέα. Και τόνισα τα σημεία που εγώ θεωρούσα ως σημεία κλειδιά. Όπως είπα και τότε, γενικά διάκυμε θετικά. Και η τροποποίηση που θα ήθελα να προτείνω ως στόχο έχει να ενισχύσει η κάθετος και να τροποποιήσει κάπως την πρόταση για να τονίσει την αποτελεσματικότητα της διοικητικής συνεργασίας ε, κατά της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής. να σας εξηγήσω σε κάπως μεγαλύτερες λεπτομέρειες τις τροποποίησεις που θέλουμε να εισαγάγουμε στο κείμενο. Πρώτα απ' όλα, ο χρονικός ορίζοντας της οδηγίας. Θα ήθελα να υπάρξει μια συγκεκριμένη μνήμα στην υφιστάμενη οικονομική κατάσταση που επισύρει μια εξαιρετική δαπάνη για την κάλυψη των αναγκών για τη χρηματοδότηση του σχεδίου ανάκαμψης και εξόδου από την κρίση. Επί τη βάση όμως της αρχής της φορολογικής ουδετερότητας και της φορολογικής ισοτιμίας ε, θα πρέπει να αποφύγουμε προβλήματα ε, φορολογικών απατών. Τώρα, επί του περιεχομένου της οδηγίας. Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογή. Το πεδίο εφαρμογή οδηγία θα πρέπει να είναι το δέον ευρύ, ούτω ώστε να συμπεριλάβει τα απαραίτητα, όλα τα απαραίτητα νομοθετικά μέσα που μπορούν να προκύψουν από μια μελλοντική φορολογική πολιτική και αρχιτεκτονική. Ούτω ώστε να μην ανοίξουμε νέες οδούς απάτης. Η ανταλλαγή ας πούμε, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτή η μορφή ανταλλαγής πληροφοριών είναι η πλέον αποτελεσματική. Ως εκ τούτου, η τροπολογία που προτείνουμε, ως στόχο έχει την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της εφαρμοσιμότητας αυτής της οδηγίας. Και θέλουμε μέσω της τροπολογίας να τονίσουμε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών με πρώτερο αίτημα κράτους μέλους θα πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικό χαρακτήρα αυτού του μέτρου για ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων. Άλλη τροπολογία. Διπλό όριο για τις πληροφορίες που ζητεί το ένα κράτος από το άλλο για μια συγκεκριμένη ε, κατηγορία συναλλασσομένων. Επίσης, προβλέπεται κατάργηση της επιτροπολογίας για τη συγκεκριμένη οδηγία. Το σύνολο λοιπόν αυτών των τροποποιήσεων που προτείνουμε για την ανταλλαγή των πληροφοριών στόχο έχει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο από το πρότυπο του ΟΣΑ που ισχύει για τις διεθνείς ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών ανά τον κόσμο. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό σύστημα που θα οδηγήσει σε μια πραγματική ολοκλήρωση. Έχουμε και άλλες τροπολογίες που προτείνουμε, ας πούμε για την έρευνα με την παρουσία υπαλλήλων αξιωματούχων από το ένα κράτος στο άλλο. η συνεργασία των φορολογικών αρχών. Εδώ βεβαίως θα πρέπει να αποφύγουμε τις συγκρούσεις μεταξύ δικαιοδοσιών και να καθορίσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας στο πλαίσιο των υφισταμένων νομοθετικών κανόνων. Επίσης, ομοίως, όπως και η ανταλλαγή πληροφοριών, ο ίδιος ο επικροτικός χαρακτήρας θα πρέπει να είναι και για τις διοικητικές έρευνες. Δηλαδή και εδώ να ισχύει υποχρέωση πληροφόρησης προς το άλλο κράτος μέλος, του τι γίνεται. Έχουμε και μια σειρά άλλων κοινών τροπολογιών ένα χρονικό ορίζοντα δηλαδή εντός του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες και μια ετήσια τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της απόρριψης αιτήματος κράτους μέλους για διοικητική συνεργασία ή για παροχή πληροφοριών. Τώρα, για την άρση του τραπεζικού απορρίτου. Η οδηγία έχει ένα περιορισμό που αφορά την φορολογική έδρα. Δεν φτάνει μέχρι την άρση του τραπεζικού απορρίτου, αλλά κάνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, στα πλαίσια όμως του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος που ισχύει σε κάθε κράτος μέλος. Θέλουμε να διαγράψουμε αυτή την αναφορά στην φορολογική έδρα, την φορολογική κατοικία και να διευρύνουμε το μέτρο αυτό σε όλο το φορολογικό τομέα σε κάθε κράτος μέλος για την άρση ομιλώ του τραπεζικού απορρίτου. Διότι ήδη κράτη-μέλη βασίζονται σε ευρύτερες διατάξεις που δεν περιορίζονται δηλαδή στη φορολογική έδρα για την άρση του απορρίτου πάντα. Ολοκληρώνω υπενθυμίζοντα αυτή η πρόταση οδηγία αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση εντάσσεται σε μια γενικότερη επιθυμία έγκριση μια κοινή στρατηγική για την ε, καταπολέμηση τη φορολογική απάτη, για τη δημιουργία μια εσωτερική ενία φορολογική αγορά και για την έγκριση των διεθνών κανόνων που θα πρέπει να διισχύουν στι διεθνεί ακριβώ συναλλαγέ. Βεβαίω υπάρχουν πολύ πιο ριζικέ διαφορές, οπότε για την καταπολέμηση της φορολογική απάτης θα πρέπει οι μηχανισμοί αυτοί ε, ανταλλαγής πληροφοριών να είναι ε, αποτελεσματικοί και να εφαρμόζονται ε, αρμονικά από όλου. Αυτά και είμαι και στην διάθεση του ή των σκιωδών εισηγητών για να συνεργαστούμε, ούτω ώστε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που θα αποστείλει στο Συμβούλιο ένα σαφέ πολιτικό μήνυμα ότι το Κοινοβούλιο είναι υπέρ μιας μεγαλύτερης φορολογικής διαφάνειας, όπως είναι εξάλλου υπέρ αυτού, πιστεύω, και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λούλινγκ. Πρόεδρε, τη της πρώτης αυτής οδηγίας που φαίνεται ότι βασίζεται σε πολύ θετικά στοιχεία και συνηθίσματα. Ε, εγώ έχω να εκφράσω κάποιες επιφυλάξεις. Ε, δεν μπορούμε να απορρίψουμε το σύνολο, αλλά βλέποντας τι διακυβεύεται, θα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετήσουμε σωστά την συζήτηση και να την κάνουμε με ευστηρότητα. Κατά γενικό κανόνα, η Επιτροπή και ο Επίτροπος Κόβατς που θα εξαφανιστεί βέβαια, αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν το τεράστιο θέμα της φοροδιαφυγής, της διαφάνειας, της ε, ε φορολογίας των ε, ε αποταμιέσεων σε μικρά μικρά κομμάτια, σαλαμοποίηση δηλαδή. Βέβαια υπάρχουν ιδιαιτερότητες για κάθε ένα θέμα, αλλά δεν πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε εις βάθος να εξετάσουμε το θέμα χωρίς να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση. Εάν εμεί ω κοινοβούλιο και αυτό εσύ και το, Γεροσυμβούλιο βέβαια δεν εξτάσουμε το θέμα παρά κατά περίπτωση, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι χρειαζόμαστε μια σφαιρική προσέγγιση, μια δέσμη δηλαδή προτάσεων. Και μόνο όταν βρεθεί μια διαιτησία πολιτική θα μπορέσουμε να νομοθετήσουμε ήρεμα. Εν τω μεταξύ, μια που όμως είμαι υποχρεωμένη, κατά κάποιο τρόπο να το κάνω, θέλω να τονίσω κάποια στιγμή που κατά τη γνώμη μου είναι προβληματικά. Όποια και αν είναι η φιλοσοφική θέση καθενός από εμά για την ανταλλαγή απόψεων, αυτόματη, κατόπιν ή αυθόρμητη, πιστεύω ότι οι συνάδελφοί μου θα με στηρίξουν σε θέματα που δεν είναι αποδεκτά. Η Κομισιόν δηλαδή να αποφασίσει με την επιτροπολογία ποιες θα είναι οι θέσεις και ποια θα είναι τα στοιχεία που θα είναι αντικείμενο της αναλύγης πληροφοριών. Αυτό θα είναι πραγματικά τελείως αβάσιμο. Ο πρώτος νομοθέτης με όλη τη διαφάνεια θα πρέπει να ορίσει το πεδίο δράσης. Ούτε είναι η Κομισιόν εκείνη η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα. Και νομίζω ότι και η συγκεντρία ακολουθεί αυτή τη γραμμή. Όσον αφορά την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ φορολογικών αρχών. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι το πρότυπο ΩΣΑ για την ανταλλαγή απόψεων και αναφέραμε εδώ στο άρθρο 26 του προτύπου σύμβαση του ΩΣΑ ή του 2002 για το Text Information Exchange Agreement έγινε δεκτό σαν ένα διεθνές πρότυπο από πολλές χώρες το Μάρτιο του 2009. Τώρα θα πρέπει να μεταφερθεί σαν κοινοτικό εκτιμένο στο ε, κοινοτικό δίκαιο. Και πραγματικά ε, απορρέει από εκεί αυτή η πρόταση του οδηγίας του, του Συμβουλίου για τη συνεργασία στα φορολογικά θέματα. Το πρώτο ποσά προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις η ζητούσα χώρα όταν υποβάλει μια αίτηση πληροφορίας θα πρέπει να καταδείξει τον ε, σημαντικό χαρακτήρα των στοιχείων που ζητάει για την περίπτωση που εξετάζει. Δεν είναι πια δυνατό στην περίπτωση αυτή η χώρα από την οποία ζητούν οι πληροφορίες να θέσει το τραπεζικό απόρριτο. και θα πρέπει όλα αυτά να ενταχθούν στην ε, οδηγία για την ε, διοικητική συνεργασία. Στην, ε, στο Λονδίνο ζητήθηκε η υπογραφή μια σειράς συμφωνιών χωρίς να ζητάει από τα κράτη-μέλη αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Θα μου πείτε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξεπερνάει τα πρότυπα του ΩΣΑ για να δώσει το καλό παράδειγμα. Εγώ απαντώ. Αυτό ήταν μεγάλο σφάλμα. Και διπλό σφάλμα. Άλλα μέρη του κόσμου προσκρούν εδώ. Γιατί το πρότυπο αυτό του δεν εφαρμόζεται παντού. Όπως το Χονγκ Κόνγκ παραδείγματος χάρη. Που το προστατεύει ο μεγάλος αδελφός, η Κίνα. Το να προχωρήσουμε περισσότερο προς το κατεύθυνση αυτή σημαίνει ότι κινούμεθα σε σφαλμένο ο, μονοπάτι. Εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να εφαρμόζουμε τα ίδια πρότυπα. Μιλούμε για ίσο πεδίο ευκαιριών για όλους. Δεύτερο σφάλμα. Η αυτόματη ανταλλαγή είναι ε, άχρηστη. Και εάν η δική οι φορολογικές αρχές έχουν αμφιβολίες δικαιολογημένες θα πρέπει μια άλλη φορολογική αρχή να απαντήσει. Αλλά αυτόματη ανταλλαγή. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Έχω το δικαίωμα ως εισηγήτρια της του να σας εξηγήσω τι εννοώ. Λοιπόν, αυτόματη ανταλλαγή όλων των στοιχείων που θα μπορούσε κανένα να φανταστεί συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση θα είχε σαν μόνο στόχο να κατακλείσει τις διοικητικές φορολογικές αρχές σε βουνά στοιχείων. Κανένας δεν θα μπορεί πια να ξαναβρει οτιδήποτε. Έχει καταδεχθεί ήδη ότι η αυτόματη ανταλλαγή απόψε που ζητάει η οδηγία για την φορολογία των αποταμιεύσεων όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί καθόλου και η Κομισιόν το παραδέχτηκε. <clears throat> Η εμπειρία είναι ξεκάθαρη. Οι φίλοι μας οι Άγγλοι κύριε ε, Πρόεδρε που τους αρέσει καταρχήν η ανταλλαγή πληροφοριών είναι εκείνοι που στην πράξη δεν την εφαρμόζουν. Δεν ανταλλάσσουν παρά αυτό που έχουν και λένε ότι δεν έχουν τίποτα σχεδόν. Απ' την άλλη, αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών, κατά τη γνώμη μου, οδηγεί σε διάφορα ρηματιματικά όσον αφορά την προστασία των ψυχίων για την ιδιωτική ζωή. Και θα ήθελα να τονίσω ότι με μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών δεν ασκούν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο, πόσο περισσότερο παραλόγω θα ήταν το συζητάμε να κάνουμε σε ένα διεθνές επίπεδο. Τέλος, η αυτόματη αυτή ανταλλαγή τίνει στο να οδηγεί σε υψηλότατο διοικητικό κόστος και όσον αφορά τους ε, οικονομικούς παράγοντες και όσον αφορά τις ε, φορολογικές δικήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί εκουσία η ανταλλαγή πληροφοριών μέσα στα πλαίσια της οδηγίας των διοικητικών πληροφοριών. Και εν αντιθέσει με αυτό που είπε η συγγήτρια, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής δεν θα πρέπει να οδηγήσει θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική χρήση. Και αυτό δεν θα γίνει με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή. Και γι' αυτό εγώ θα ήθελα να πω ότι είμαι αντίθετη στην ύπαρξη εκπροσώπων ενό κράτου μέλου στι ε, φορολογικέ διοικήσει μια άλλη χώρα μέλου. Αυτό καταπατά την ε, ανεξαρτησία κάθε κράτου. Ε, και τότε κάθε κράτο θα πρέπει να δυσπιστεί έναντι οποιοδήποτε άλλο. Αυτή όμως η γενικευμένη δυσπιστία είναι απαράδεκτη. Γιατί να μην στείλουμε τότε κατευθείαν στρατό. Uh, Κοιτάξτε, είχαμε πει ε, να μιλήσετε για 10 λεπτά. Τελικά μιλήσετε 3 λεπτά παραπάνω από τον εισηγητή. Δεν μπορεί να μιλήσει τόσο πολύ ο κάθε ο εισηγητής. Ε, βέβαια, ε, ξέρω ότι διαφωνείτε με τους άλλους ε, και γι' αυτό σας άφησα, αλλά εν πάση ελπίζω οι υπόλοιποι εισηγητές να είναι λίγο πιο σύντομοι. Μήπως, μπορεί τώρα, μήπως μπορείτε να προβλέψετε χρόνο και για την Κομισιόν, γιατί εγώ θα ήθελα να γνωρίζω την άποψη της Κομισιόν. Εντάξει, αλλά έχω ένα χρονοδιάγραμμα και η κυρία Λούλινγκ μου το έκανε άνω κάτω. Ο κύριος Λάμπερτ, κοιτάξτε, εγώ δεν θα μιλήσω για 10 λεπτά να είστε σίγουρος. Εδώ κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ φίλων. Αλλά εδώ μιλάμε για φίλους, μιλάμε για χρήμα. Κοινοτικό χρήμα, κυρία Λούλινγκ. Οπότε δεν είναι και τόσο δευτερεύον το ζήτημα. Ξέρετε πόσο κοστίζει η φορολογική απάτη. Ξέρετε το δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών μελών λόγω της φοροδιαφυγής και της απάτης. Είναι και, η ώρα λοιπόν να πειράσουμε σε μια άλλη ταχύτητα. Ανώτερη. Όταν λέτε εσείς χαλάρωση, εσείς χαλάρωση των κανόνων, ουσιαστικά λέτε φορολογικό βάρος προς τον τίμιο πολίτη που πληρώνει το φόρο του. Κυρία Λούλινγκ, σας παρακαλώ, εγώ δεν σας διακόψα, μη με διακόπτετε. Και ξέρουμε και από πού κατάγεστε, έτσι, ποια είναι η χώρα σας. Οπότε θα ήθελα να πω ότι εμείς ως πράσινοι υποστηρίζουμε την έκθεση Άλβαρεθ και σας συγχαίρω κύριε Άλβαρεθ για το έργο σας. Θα ήθελα υπό αυτή την έννοια να διαφωνήσω και με την κυρία Λούλινγκ. Ο ΩΣΑ δεν είναι το χρυσούν πρότυπο ούτε από πλευρά δημοσιονομικών, ούτε από πλευρά φορολογική αποτελεσματικότητα. Γιατί η αποτελεσματικότητα είναι το ζητούμενο και πιστεύουμε ότι η αυτόματη ανταλλαγή θα πρέπει να είναι ο κανόνας. Και μην ανησυχείτε κυρία Λούλινγκ, γεννηθήκατε κατά πάσα πιθανότητα πριν την τεχνολογική επανάσταση. Και πλέον δεν τίθεται θέμα αφού είναι αυτόματη η ανταλλαγή πληροφοριών, το μηχάνημα το αναλαμβάνει. Ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτα. Απλώς μπορούμε να ανοιχνεύουμε αυτούς που προβαίνουν σε απάτες. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι αυτή η αντιπαραβολή και αντιπαλότητα μεταξύ επιτροπολογίας και συγκεκριμένου καταλόγου ε, μου δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί αν κάτι ξεχάσουμε να βάλουμε στη λίστα, αν προκρίνουμε τη λύση της λίστας και ξεχάσουμε κάτι να βάλουμε στη λίστα, αυτό σημαίνει παραθυράκι. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λάμπερτ. Επόμενος ομιλητής. Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση γίνεται ιδιαίτερα παθητική, δείχνει πάθος, ευχάριστο αυτό και γι' αυτό και εγώ θα χρησιμοποιήσω τη δική μου τη μητρική γλώσσα για να παραμείνω στο ύφος αυτό της συζήτηση. Να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να φερθώ στο ότι ο αγώνας κατά της ε, φοροαπάτης είναι πολύ σημαντικός. Κανείς από εμά δεν αμφισβητεί ότι είναι σημαντικό να ε, καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή και την φοροαπηφογή. Η κυρία Λούλινγκ, εξ όσων γνωρίζω, έχει δίκιο σε αυτά που είπε. Αν δηλαδή επρόκειτο να συζητήσουμε για ένα πραγματικό αγώνα κατά της φοροδιαφυγής, ε, θα έπρεπε να αναφερθούμε στην διαφάνεια των συστημάτων. Η φόροι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο περίπλοκοι, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τόσο εξαιρέσεις ως προς το ΦΠΑ, γιατί όσο πιο πολλές εξαιρέσεις υφίστανται, τόσο πολύ πιο εύκολο καθίσταται να ε, προκύψουν περιπτώσεις ε, φοροδιαφυγής. Τέλος, να σας πω ότι εγώ δεν συμφωνώ με την έννοια ότι η οικονομική ύφεση θα δικαιολογεί οποιαδήποτε ε, παρέμβαση στην οικονομία μιας χώρας και στο φορολογικό σύστημα μιας χώρας. Εγώ πιστεύω ότι οι νομοθέτες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσον αφορά αυτό το σημείο. Η ε, τρίτη μου παρατήρηση αφορά αυτά που είπε η κυρία Λούλινγκ και πάλι συμφωνώ μαζί της. Εγώ θέλω να σας πω ότι το τρίτο δικό μου σημείο αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών. Αν λοιπόν η ανταλλαγή πληροφοριών γίνει δεσμευτική, τότε ε, θα είναι πολύ πιο εύκολο να ρυθμίζονται διαφωνίες ανάμεσα στις φορολογικές αρχές, πολλές φορές μάλιστα και περιτές. Ε, βεβαίως εμείς είμαστε υπέρ του να δίδονται πληροφορίες οποτεδήποτε ζητούνται και όχι αυτόματα. Τελευταίο μου σημείο και τέταρτο θα ήθελα να μου επιτρέψετε να φέρω ένα παράδειγμα δεν νομίζω ότι αυτό που θα πω έχει σχέση με τη δική μας την Επιτροπή, έχει περισσότερο με την Επιτροπή Βιομηχανίας σχέση, αλλά το δώσει είναι ενδεικτικό το παράδειγμα. Ε, μία μεγάλη ε, εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της Τσεχίας έχει δεχθεί την έρευνα από τις Βρυξέλλες πάρα πολλοί υπάλληλοι των Βρυξελών πήγαν σε αυτή, στον οργανισμό για να ψάξουν τα στοιχεία τους. Το ίδιο συνέβη και στην Πράγα και τους υπολογιστές και τα πάντα. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος. Το θέμα είναι κατά πόσον η παρουσία ξένων ελεγκτών και ξένων υπαλλήλων είναι πάντα σωστή ή όχι. Με τον τρόπο αυτό ανοίγουμε ένα πολύ επικίνδυνο δρόμο. Έχουμε μία μεγάλη δέκο, μία εταιρεία κοινή ωφελία που συμμετέχει σε διαγωνισμό, δημόσιο διαγωνισμό για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού, άρα δηλαδή οποιαδήποτε διαρροή πληροφορίας μπορεί να είναι πολύ σημαντική για αυτήν την εταιρεία. Εγώ πιστεύω ότι οι κανόνες πρέπει να είναι σαφείς, και πρέπει να είναι επίση σαφές το ποιος αποφασίζει τελικά. Οι ε, εθνική εθνικοί υπάλληλοι ή οι ξένοι που έρχονται και τους επισκέπτονται. Και εγώ, με συγχωρείτε να σας πω, να σα ενημερώσω, και εγώ γεννήθηκα πριν από την ε, τεχνολογική επανάσταση. Για να το ξέρετε απλά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, αυτό το σύστημα των ελέγχων, αυτό πρέπει να προσαρμόζεται στην αγορά. Τώρα λοιπόν έχουμε μια ε, πολύ μεγάλη κοινή αγορά όπου τα συστήματα είναι ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι ανάλογο και το σύστημα ελέγχου. Πρέπει όμως να είμαστε και πολύ προσεκτικοί. Παραδείγματο χάρη, αν ε, τελικά το Κοινοβούλιο ζητήσει η ανταλλαγή δεδομένων να γίνεται με πολύ μεγάλη σύνεση και αν πράγματι μας ενδιαφέρει η προστασία των δεδομένων, γιατί αυτό είναι κάτι που αφορά τους πολίτες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, εγώ όλα αυτά τα βρίσκω σωστά. Όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύονται και σε περιπτώσεις φορολογικών διενέξεων. Το να έρεται το τραπεζικό απόρριτο, αυτό είναι κάτι διαφορετικό από το να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, για να αρθεί το απόρριτο πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλές εγγύησεις. Ε, το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν πρέπει να γίνονται όλα αυτόματα. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο πράγματι υφίστανται οι απαραίτητε εγγύσει για την ανταλλαγή πληροφοριών. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν υπάρχουν ε, κάποιες ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά, τότε η ανταλλαγή πληροφοριών θα ήταν καλύτερα να γίνει μέσα από σχετικό αίτημα. Εγώ το προτιμώ αυτό. Για μένα είναι καλύτερη λύση. Κοιτάξτε, σας υποσχέθηκα ότι θα είμαι σύντομη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Άλβαρεθ για την πολύ καλή δουλειά της. Εξάντλησα τα ισπανικά μου και περνάω τώρα στα Ουγγρικά. Είναι όντως απαραίτητο να εμβαθύνουμε επί του προβλήματος και να δούμε τι ακριβώς γίνεται, πόσα προβλήματα και πόσα χρήματα υπάρχουν και στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την πρόταση και εγώ την ίδια άγουσα θα λάμβανα με την κυρία Άλβαρεθ. Στην αρχή δεν καταλάβαινα γιατί θα πρέπει να υπάρχουν δύο όρια. Τώρα όμως το κατάλαβα πολύ καλύτερα και συμφωνώ αναείδος εισοδήματος και ένα όριο τιμής, ανώτατης τιμής. Αν κατάλαβα καλά, αυτό είναι το διπλό όριο. Και νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Επίσης συμφωνώ και με τις τροποποιήσεις, με τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν Όντως, η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μια αντιπαλότητα και σε έναν ανταγωνισμό για το ποιο είναι ο αρμόδιος για το τάδε και ποιο είναι ο αρμόδιος για το δίνα. Το ζητούμενο είναι η συνεργασία και η αποτελεσματικότητα. Επίσης, σύμφωνο με το ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο κείμενο για να καθορίσουμε ε, το αντικείμενο της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το αφήσουμε ε, όμοιρο της επιτροπολογίας. Δηλαδή δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί μέσω επιτροπολογίας αλλά μέσω νομοθετικών ε, προτάσεων. Τώρα, για τα τελωνία υπάρχει ήδη συνεργασία ας πούμε. δεν συμφωνώ ότι θα πρέπει να συμπληθούν εδώ στον κατάλογο τα τελωνία. Πάντως υποστηρίζουμε την εργασία της ε, εισηγήτριας και τις ε, τροποποιήσεις που η ίδια πρότεινε. Ευχαριστώ. Thank you. Um, uh, we have a slight problem there with the, the translation. Mr. Bullman, very, very briefly, because I would like to... Κύριε Μπούλμαν, πολύ γρήγορα γιατί θα ήθελα να δώσω το λόγο και στην Κομισιόν. Ναι. Κοιτάξτε, ε... <clears throat> εγώ δεν θα καταχρηστώ τους χρόνου, εγώ θέλω να αναφερθώ στους αδέλφους που <laughs> εξάπτωται η συζήτηση, άσχετα από το καν γεννήθηκαν πριν ή μετά την τεχνολογική επανάσταση, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι η εξασφάλιση των φόρων για τα κράτη-μέλη είναι ένα βασικό αγαθό και θα πρέπει βέβαια στους σύγχρονους καιρούς να α, χρησιμοποιούμε σύγχρονα μέσα και γι' αυτό θα ήθελα να ακολουθούμε την έκκληση της ε, συναδέλφου Αλφαρέας να συνεργαστούμε και να μην παρεμποδίζουμε. Πρέπει σαν κοινοβούλιο να μιλάμε με μία φωνή. Ευχαριστώ. Okay, um, from, from, from... Ωραία. Από την Κομισιόν, ο κ. Ναπών έχει το λόγο. Bien, merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κάποιες σύντομες ε, παρατηρήσεις. Κυρία Λούλινγκ, δεν είναι ο κύριος Κόβατς ο επίτροπος που εγκρίνει τις προτάσεις. Το σώμα των επιτρόπων εγκρίνει την οποιαδήποτε πρόταση. Είναι συλλογικό όργανο. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, έχουμε μια συντονισμένη στρατηγική. Σε τέτοιο βαθμό που σήμερα συζητούμε δύο θέματα της διοικητικής συνεργασίας και αύριο το πρωί ένα τρίτο. Οπότε είναι μια συντονισμένη προσέγγιση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εις ό,τι αφορά τώρα την ιδιαιτερότητα της ε, κοινότητας, ε, η ιδιαιτερότητα αυτή είναι η εσωτερική αγορά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Κομισιόν προστεύει ότι θα πρέπει να πάμε πέρα από τα διεθνή πρότυπα του ΟΟΣΑ. Ο ΟΟΣΑ διεθνέ επίπεδο δεν αφορά την εσωτερική αγορά. Δεν υπήρχε εσωτερική αγορά για τον ΟΟΣΑ. Είναι ένας ελάχιστος κοινός αλλά στην κοινότητα θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Τώρα, να λέμε ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών δεν ισχύει για τις αποταμιεύσεις είναι λάθος. Είναι λάθος. Λειτουργεί και λειτουργεί τέλεια. Σε τέτοιο βαθμό που το Λουξεμβούργο που κάνει κράτηση, παρακράτηση στην πηγή ανταλλάσσει δύο εκατομμύρια φακέλους για εθελούσιες δηλώσεις. Ακόμα και στο Λουξεμβούργο γίνονται εθελούσιες δηλώσεις. Και όπως είπε ένας βουλευτής, εφόσον υπάρχει η τεχνολογία θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Τα κράτη-μέλη είναι σε θέση να την αξιοποιήσουν. Ίσως ό,τι αφορά τώρα την ανταλλαγή πληροφοριών μετά από αίτημα και όχι την αυτόματη δηλαδή. Όντως, όντως οι συνθήκες είναι τέτοιες που είναι πολύ δύσκολο να ισχύσει αυτό το μέτρο της ανταλλαγής πληροφοριών μετά από έτοιμα. Γιατί? διότι απλούστατα καλείστε να δώσετε έναν αριθμό πληροφοριών εάν τις κατέχετε. Η φορολογική αρχή του κράτους μέλους που το ζητεί θα μπορούσε από μόνη της να συλλέξει πιο αποτελεσματικά το φόρο. Προκειμένου περί άλλων μέτρων για την επιτόπου παρουσία υπαλλήλων άλλου κράτους μέλους. Αφού υπάρχει για το ΦΠΑ, γιατί να υπάρχει πρόβλημα εδώ σε θέματα άμεση ε, φορολογία. Για την προστασία των δεδομένων συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Πολύ λεπτό και σημαντικό ζήτημα για το ΦΠΑ, α πούμε, για το ΦΠΑ. Εμείς ε, ήρθαμε σε επαφή με τον Ευρωπαίο Επόπτη, τον υπεύθυνο για την ε, προστασία των δεδομένων. Το Κοινοβούλιο έλαβε αντίτυπο τη της του οργάνου αυτού που λέει σαφώ ότι το μοντέλο του ΦΠΑ μπορεί να ισχύσει και στην άμεση φορολογία. Και εμείς λέμε ότι πληρούνται τα κριτήρια για την προστασία των δεδομένων. Βεβαίως ο επόπτης ζήτησε από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο να επιφέρει κάποιες διευκρινήσεις και να εγγυηθεί το απόλυτο απόρριτο εις ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Και νομίζω ότι τα κράτη-μέλη είναι πολύ προσεκτικά επ' αυτού. Σε τέτοιο βαθμό που απέκλεισαν την Κομισιόν από οποιαδήποτε δυνατότητα πρόσβαση σε αυτές τι πληροφορίες. Η Κομισιόν βρίσκεται μόνο εδώ για να διαχειριστεί ηλεκτρονικά αυτές ε, τις ανταλλαγέ πληροφοριών, αλλά πρόσβαση στο περιεχόμενο των πληροφοριών δεν έχει και ούτε θα έχει. Αυτά. Και βεβαίω να δηλώσω την πλήρη ικανοποίηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεση Άλβαρεθ και τι τροπολογίε. Κυρία Άλβαρεθ, παρακαλώ, εάν θέλετε να συγκεφαλαιώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτη μου έκθεση ήταν. Και ποτέ δεν φανταζόμουν ότι αυτό θα ήταν το θέμα της πρώτης μου εκθέσεως διοικητική συνεργασία για φορολογικά θέματα. Και εξεπλάγιν. Εξεπλάγιν. Που είδα ότι η συνεργασία ανέβαινε κρεσέντο που λέμε και ενισχυόταν κάθε φορά όλο και περισσότερο. Ευτυχές, ευτυχέστατο ολοκλήρωσα αυτή τη σύντομη σκέψη. Δεύτερον, φαντάζομαι ότι συμφωνούμε ότι ισχύει η εθνική κυριαρχία, εις ό,τι αφορά τα φορολογικά θέματα. Χωρίς όμως τις κατάλληλες πληροφορίες δεν μπορεί το κράτος μέλος να εφαρμόσει τη φορολογική του πολιτική. Δηλαδή είναι απαραίτητη η ανταλλαγή πληροφοριών για την άσκηση της εθνικής φορολογικής κυριαρχίας. Επαναλαμβάνω για να εφαρμόσει τη φορολογική του πολιτική, ένα κράτος μέλος χρειάζεται πληροφορίες που κατέχει άλλο κράτος μέλος. Και μην ξεχνάτε ότι στο κάτω-κάτω της γραφής μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την Ιορδανία, το Χονγκ Κόνγκ ή τη Σιγκαπούρη. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για μια ομάδα χωρών των πλέον ανεπτυγμένων χωρών που θέλουν να προχωρήσουν για να βρουν μια λύση που δεν μπορούν να βρουν μόνα τους τα κρατήμελη. Γι' αυτό μιλάμε. Προσπαθούμε να πορευθούμε λοιπόν μαζί. Τώρα, από τον κύριο Στρέκ και ζητώ συγγνώμη αν δεν προφέρω σωστά το επώνυμό του. που λέει ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε στα χωράφια τη εθνική κυριαρχία των κρατών μελών και το συνδέω αυτό με το προηγούμενο. Ζητώ συγγνώμη αν έδωσα αυτή την εντύπωση και ε, πραγματικά δεν ήθελα να το πω αυτό. Εγώ είπα ότι στην οδηγία καλό θα ήταν να αναφέρεται ότι ο πολίτης στη στιγμή κρίσης να έχει τη δυνατότητα να πει, να αναγνωρίσει στο δημόσιο, στην πολιτεία το γεγονός ότι παραμβαίνει για να πατάξει την φορολογική απάτη. Ποτέ δεν είναι αποδεκτή η φορολογική απάτη, αλλά είναι ακόμα λιγότερο αποδεκτή σε στιγμές κρίσης. Δεν πρόκειται λοιπόν για παρεμβατισμό. Κυρία Λούλινγκ είναι αυτή που έθεσε τα πιο σημαντικά προβλήματα και θα τα πω γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Η γενική προσέγγιση Μάλλον, να το πω αλλιώς, ε, αυτή είναι μια ειδική περίπτωση που εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Έτσι, μιλάω για την ανταλλαγή πληροφοριών. Εδώ μιλάμε για την καταπολέμηση τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή. Μην το ξεχνάμε. Δεν μιλάμε για γενίκευση αυτού του α, μέτρου. Και είπε κάποιο συνάδελφο ότι αν κάνουμε μια λίστα, αν ξεχάσουμε κάτι και μείνει εκτό λίστα, ανοίγει το παραθυράκι προ την απάτη. Σωστό. Τέλος, στην κυρία Λούλινγκ θα ήθελα να πω μάλλον είπε η κυρία Λούλινγκ ότι δεν θα ωφελήσει κανέναν αυτή η οδηγία. Έτσι το απατέ. Συγγνώμη κυρία Λούλινγκ, αλλά πιστεύω ότι απατάστε. Ότι πλανάστε. Πλάνιν ικτράν. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε την πόρτα ανοιχτή στους απατεώνες. Να έχω εγώ ως κράτος μέλος μια πληροφορία που ξέρω ότι θα βοηθήσει άλλο κράτος μέλος να εφαρμόσει πιο αποτελεσματικά φορολογικά μέτρα και να καταπολεμήσει την απάτη είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Αυτά και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που μου έδωσαν ιδέες. Αυτό το διπλό όριο εσείς ήσασταν κυρία Λούλινγκ που μου το προτείνατε την τελευταία φορά. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους σκιώδεις οι συγκεκριτές που μου έδωσαν ιδέες για να καλύψω θέματα τα οποία είχα ε, ξεχάσει. Και κυρία Λούλινγκ, μπορείτε να είστε ήσυχοι γιατί πιστεύω ότι δεν θα είναι δαπανηρό το μέτρο και θα είναι επωφελές για όλους τους πολίτες με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο συγκητής για την επόμενη έκθεση είπε ότι δεν θα μακρηγορήσει ιδιαίτερα και αυτό σας άφησα να μιλήσετε κάπως παραπάνω. Περνάμε τώρα στην αμοιβαία συνδρομή για την ίσπραση απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δοσμούς και άλλα μέτρα και την εξέταση σχεδίου γνωμοδότηση από τον κύριο Στόλογιάν. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι πραγματικά πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το σχέδιο οδηγίας που θέλει να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της ε, ίσπραξης απαιτήσεων από φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα είναι απαραίτητο μέτρο. Γιατί αυτή τη στιγμή η αποτελεσματικότητα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Είχαμε μία ανταλλαγή απόψεων για την πρώτη αυτή οδηγίας και είπα ότι ένα από τα συζητήσιμα θέματα που αναφέρεται στην προηγούμενη έκθεση επίσης ήταν το γεγονός ότι η αποδοχή της παρουσίας υπαλλήλων των φορολογικών αρχών ενός κράτους μέλους σε ένα άλλο κράτος μέλος είναι απαραίτητη. Σε αυτή εδώ την πρώτη οδηγία όμως η δυνατότητα αυτή αναφέρεται μόνο με συμφωνία των δύο μερών. Αν τα δύο μέρη δηλαδή συμφωνούν και πληρούν οι προποθέσει ούτω ώστε να εκπρόσωπος φορολογικών αρχών από τη μία χώρα μέλος να είναι παρόν σε μια άλλη χώρα, είναι εντάξει. Οι δύο χώρες αυτές μεταξύ τους δηλαδή θα δεχθούν ή δεν θα δεχθούν αναλόγως αυτή την παρουσία. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να πω ότι έχω μία μόνη τροπολογία η οποία διευκρινίζει το ότι όταν υπάρχουν έγγραφα που παρατούνται αυτά θα πρέπει να είναι ε, δυνατότητα να στέλνουν όχι μόνο τα πρωτότυπα αλλά και επιστοποιημένα αντίγραφα. Πρόεδρος, μπορούν οι σκιώδεις ηγητές να σχολιάσουν παρακαλώ. Okay. Oui, comme Ναι, είμαι σκιώδης ηγητής για την ε, σοσιαλιστική και δημοκρατική ομάδα. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Όπως είπα ήδη στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων, νομίζω ότι ο εισηγητής τόλισε στο έγγραφο αυτό τις κύριες αδυναμίες του κειμένου που υποβάλλει η Κομισιόν. Η ομάδα μου και εγώ προσωπικά ήμασταν κάπως απογοητευμένοι γιατί η έκθεση που μας παρουσιάζεται σήμερα είναι πάρα πολύ σύντομη. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα κάνουμε καλά να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες, ιδίως όσον αφορά τις προθεσμίες, όσον αφορά τα κατόφλια και όσον αφορά τις υποχρεώσεις που εμπίπτουν στη χώρα που ζητά συνεργασία για την ανταλλαγή απόψεων. Ελπίζω να μην φανεί αυτό στην κυρία Λούλη. Δεν αφιβάλλω ότι βάσει των τροπολογιών αυτών θα μπορέσουμε να βρούμε ισχυρές βαστικές λύσεις για να μπορέσουμε έτσι να αυξήσουμε η δυνατότητα των κρατών μελών να αποκτήσουν από τους ε, πολίτες ε, το σεβασμό των φορολογικών των υποχρεώσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αν κάποιος από την άλλη μήπως θέλει να σχολιάσει. Ashley Fox. Uh, Mr. Jürgen Uh, um, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά βάση μπορώ να συμφωνήσω με την πρόταση. Δεν θα μόνο να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα σημείο. Και σχετικά θα υποβάλω και μια σχετική τροπολογία. Χρειάζεται να προετοιμάσουμε μια μελέτη για το διατεκτικό τομέα στο τομέα της φορολογίας. Θα ήταν καλό να ξέρουμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν στα 27 κράτη-μέλη όσον αφορά παραδείγματο χάρη τα μητρώα των ακινήτων, ποια είναι τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί σε τράπεζα δεδομένου για το θέμα αυτό. και επίσης και τι προθεσμίες ισχύουν. Αν είχαμε μια συγκριτική μελέτη θα μπορούσαμε νομίζω να την ε, παρουσιάσουμε στα κράτη-μέλη προς όφελος όλων γιατί θα γινόταν πιο εύκολα η ανταλλαγή των στοιχείων και θα ξέραμε τι λειτουργεί σε ποια χώρα, τι δεν λειτουργεί. Θα ήταν πάρα θετικό αυτό νομίζω. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν θέλει κάτι να πει. Όχι, Πρόεδρε. Απλώς όμως ήθελα να σας δώσω μια πληροφορία όσον αφορά τη συμβολή για την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό απεσύρθη μετά τις συζητήσει στο Συμβούλιο από την πρώτη οδηγία, γιατί όταν είχαμε υποβάλει εμεί την πρόταση, ο κατανοησμός που είχε υποβάλει ο συνάδελφος Ζωντών δεν είχε ακόμη υιοθετηθεί. Τώρα υιοθετήθηκε υιοθετήθηκε συγγνώμη, και θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Μαΐου 2010, οπότε θα είχαμε επικαλύψεις μεταξύ αυτής της οδηγίας και των κανονισμού που υιοθετήθηκε. Γι' αυτό το λόγο αυτό το θέμα δεν τίθεται πια σήμερα. Κατά τα άλλα δεν έχω κανένα σχόλιο να κάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής. Ε, πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους τους αδέλφους για τα σχόλιά τους και φυσικά θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει και μια προθεσμία για τις ε, 10 Δεκεμβρίου νομίζω. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Καταφέραμε να αρχίσουμε και 10 λεπτά νωρίτερα. Ο εισηγητής για το επόμενο θέμα δεν είναι ακόμα παρόν. Οπότε θα διακόψουμε και στις 5 θα συνεχίσουμε, θα έχει έρθει και ο Ζων Πολ. Okay, can everybody start to sit down, please? Thank you. If we if we calm ourselves down um, for what, I, what, what, what might be another sparkling session. Κοιτάξτε, ε, καθίστε στις θέσεις σας παρακαλώ να συνεχίσουμε. Um, λοιπόν, πάμε στο σημείο υπαριθμών 7 της ημερήσιας διάταξης που είναι η οδηγία για τους διαχειριστές εναλλακτικών επενδύσεων. Έχουμε λοιπόν το σχέδιο της έκθεσης του εισηγητή και ως εκ τούτου θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Ζαν Πολ για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συναδελφοί, αυτή η έκθεση αναμένεται φαίνεται καυτά. Πολλοί ήρθαν να μου εξηγήσουν ότι ήταν καλή οδηγία. Αλλά εάν δεν προσθέσουμε πολλά θα ήταν ακόμη καλύτερη. Εμένα η πρότασή μου προφανώς είναι να τη διατηρήσουμε την οδηγία αυτή με το πεδίο εφαρμογή τη και εν να ενδυναμώσουμε τον διαγωνισμό που προβλέπει η Κομισιόν. Είχα ήδη την ευκαιρία να σας πω ότι αυτή η έκθεση αποτελεί μια βάση εργασίας και δεν είναι προφανές ένα τελειοποιημένο έγγραφο, αλλά αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα συζήτηση μεταξύ μας. Εγώ θα ήθελα να μην επισέλθω στις λεπτομέρειες ούτως ώστε η συζήτηση να γίνει γύρω από τα κύρια θέματα της οδηγίας. Και όταν συμφωνήσουμε πάνω στις γενικές γραμμές, ή άμα τις τροποποιήσουμε κιόλας, τότε μπορούμε να μπούμε στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε τις δυνατότητες να υποβάλλετε τροπολογίες που θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να συζητήσουμε και θα μας επιτρέψουν να δώσουμε μορφή στην πρόταση αυτή της οδηγίας πριν να περάσουμε σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Τα κύρια στοιχεία. Και θα σας πω καταρχήν ότι το πεδίο εφαρμογής παραμένει αυτό που είχε ε, προβλεφτεί. Όλα δηλαδή εκτός από την δικαιοσύνη. Εγώ διάγραψα τα κατόφλια γιατί ξέρω ότι όταν υπάρχουν κατόφλια υπάρχουν επιπτώσεις των κατοφλίων δηλαδή η δημιουργικότητα των ε, οικονομολόγων και των νομικών ε, κάνει να αναζητήσουν ε, δυνατότητες να ξεπεράσουν τις οδηγίες και από την άλλη μεριά θέλω να υπάρχει μια αρχή αναλογικότητας ότι διαχείριση για τις μικρές επιχειρήσεις να λαμβάνει υπόψη το πραγματικό τους μέγεθος για να μην τους επιβάλλει υπερβολικούς ε, κανόνες. Αυτή μετά εξέτασα το θέμα των ε, τρίτων χωρών. Τι θα γίνει δηλαδή με εκείνα, τα, εκείνους τους οργανισμούς επενδύσεων που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν θα πω στις λεπτομέρειες, αλλά θα σας πω ότι η βασική ε, πρόταση είναι ότι θα πρέπει να είναι ένα φρούριο η Ευρώπη και να αγνοεί τι γίνεται γύρω τη, από την άλλη μεριά θα πρέπει να είναι και σουρωτήρι. Και ό,τι όλοι οι κανόνες που εφαρμόζονται να μην έχουν καμία αποτελεσματικότητα λόγω διατάξεων που θα ανάξουν διάπλετες πόρτες ε, της ε, Ευρώπης σε διαχειριστές οργανισμών επενδύσεων που δεν είναι διαγωνισμένοι. Γι' αυτό θα έλεγα το Ευρωπαϊκό ε, Διαβητήριο να δοθεί όπως ειδικές τράπεζες σε εκείνους τους συγκεκριμένους διαχειριστές μιας, ε, από μια χώρα μέρες Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη για μια μεταβατική περίοδο να προβλέψουμε ιδιωτικές επενδύσεις που δίνει τη δυνατότητα μιας επίλυσης. Και λέω για μεταβατική περίοδο, γιατί προφανώς το ιδανικό θα ήταν να έχουμε εναρμονισμένο διαγωνισμό στον τομέα αυτό. Φοβούμε όμως ότι αυτή τη στιγμή η ιδέα αυτή της εναρμόνισης, αναγνώριση ισοτιμίας κλπ. θα είναι μάλλον μη ρεαλιστική και δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί αμέσως. Γι' αυτό προτείνω να διατηρηθεί η ιδιωτική επένδυση ανοίγοντα τις ε, προοπτικές για καλύτερο ευρωπαϊκό διακανονισμό τα επόμενα χρόνια. Ετέθη επίση το θέμα του καταθέτη, της ευθύνη αυτού. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Εγώ λέω ότι όσο πάει υπάρχουν και λιγότεροι υποψήφοι γι' αυτό, γιατί αυτό το επάγγελμα δεν είναι πια τόσο αποδοτικό και ε, ενέχεται πια πολύ μεγάλη ευθύνη. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε οι ευθύνε του να, διακανε... να ορίζονται ξεκάθαρα και να μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους που ε, δικαιολογούν, την ε, ευθύνη του. Το θέμα του, της ε, του φαινομένου μοχλού Είναι σημαντικό. Θα πρέπει να εξασθεί με στα πλαίσια της αξιολόγησης των ιδίων ε, κεφαλαίων της ε, τράπεζας, γιατί οι τράπεζες θα προβλέπουν έναν έλεγχο αυτού του φαινομένου μοχλού. Δεν υπάρχει όμως κανένα μαγικός αριθμός να πούμε δηλαδή το ιδανικό μου είναι 2, 3, 5 ή 10 και η Κομισιόν όταν λέει ότι θα πρέπει να υιοθετήσει τα απαραίτητα μέτρα παρουσιάζει μια καλή λύση γιατί αυτό θα είναι πάρα πολύ αργά. Προτείνω λοιπόν μια ρεαλιστική λύση και θα έλεγα ότι ο επόπτης και εγώ τοποθετήθηκα μέσα στην νέα προοπτική του Ευρωπαίου επόπτη που προετοιμάζω το σχετικά κείμενα αυτή τη στιγμή θα πρέπει πλέον να ελέγχει ο επόπτης σε δύο στάδια. Καταρχήν τη στιγμή κατά την οποία ο διαχειριστής των ε, πόρων αυτών υποβάλλει τις πληροφορίες στην διακτονιστική υπηρεσία θα πρέπει να αναφέρει ποια πολιτική θέλει να ακολουθήσει όσον αφορά το φαινόμενο μοχλού και εκείνη τη στιγμή ο Βεπόπ θα πρέπει να μπορεί να αξιολογήσει κατά πόσο η πολιτική αυτή είναι διψοκίνδυνη ή όχι. Κατά δεύτερον, καθ' όλη τη διάρκεια ζωή ε, του οργανισμού επένδυση θα πρέπει ο Επόπτη να ελέγχει κατά πόσον η πολιτική που προαναγγέλει ο διαχειριστή ακολουθείται ή αποκλίνει από εκείνο που είχε προαναγγείλει. Στην περίπτωση αυτή θα μπορεί ο Επόπτη να ελεγχει κατα ποσον η πολιτικη που προαναγγελει ο διαχειριστη ακολουθειται η αποκλινει απο εκεινο που ειχε προαναγγειλει στην περιπτωση αυτη θα μπορει ο εποπτης να προειδοποιησει τον ε, διαχειριστή ή να δώσει ας πούμε και μια προειδοποίηση ώστε οι επενδυτές να δούνε πόσο κίνδυνο διατρέχουν. Και όταν είναι πάρα πολύ σοβαρές περιπτώσεις θα μπορεί η Κομισιόν ή ποιος άλλος να περιορίσει το φαινόμενο αυτό του μουχλού. Αξιολογητής. Η Κομισιόν αναφέρθηκε σε έναν ανεξάρτητο αξιολογητή στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι εκείνοι που μπορούν να αξιολογήσουν έναν οργανισμό επένδυσης που ίσως δεν χρειάζεται καν σε private equity Οι καταθέτες και οι επόπτες θα μπορούν να τα κάνουν. Γι' αυτό να διαγράψουμε αυτή την αφορά στην ανεξαρτησία. Εθνικά όποιος θέλει να έχει έναν ανεξάρτητο αξιολογητή μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει όμως να υπάρχει στην, ε, ε στον οργανισμό διαχείρισης ε, μέτρα που να αποφεύγουν τη σύγκρουση συμφερόντων. Αναφέρομαι επίσης στο θέμα της πληρωμής των διευθυνόντων. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα θα πρέπει να προσανατολιστεί στους κανόνες που υπάρχουν για την, ε, <clears throat> για την πληρωμή, για την χορήγηση δανείων. Μία πλαισίωση θα πρέπει να είναι δυνατή όταν χρειάζεται και θα πρέπει να γίνεται για να απευθεί ο συστημικός ε, ε, κίνδυνος. Όσον αφορά του επενδυωμένου κεφαλαίου, νομίζω ότι η οδηγία που παρουσιάζει μια κοινή δέσμη μέτρων είναι ανεπαρκής και θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να λεφθεί υπόψη ποιες ιδιαιτερότητες έχει το επενδυτικό κεφάλαιο για να μπορέσουν να περιοριστούν τυπικότητες όταν δεν χρειάζονται ή όταν δεν υπάρχει ο κίνδυνος. Γιατί τα κεφάλαια επένδυσης είναι ε, ε, δεσμεύσεις διαρκείας με μία διαχείριση και πληρωμή που επιστρέφει στους επενδυτές και απορρέει από την ίδια την αγορά. Έτσι θα μπορούμε νομίζω όσον αφορά το επενδυόμενο κεφάλαιο να περιορίσουμε τις τυπικότητες στο απαραίτητο. Αναφέρθηκα στην εποπτεία όσον αφορά τις αρμοδιότητες των κρατών μελών θα πρέπει και εδώ νομίζω να συνδυάσουμε στα πλαίσια της νέας αρχιτεκτονικής ε, της ισχύς ε, των αρχικών χωρών προέλευσης ε, της χώρας προέλευσης και της τρέχουσας χώρας υποδοχής υπάρχει και το θέμα της, ε, ε της ε, συνεργίας με άλλα κείμενα, όπως M και λοιπά. Να, προσπάθησα να λάβω υπόψη τα κείμενα αυτό και όπου ήταν δυνατόν αναφέρθηκα στους όρους των οδηγιών αυτών όταν ε, πρόκειται για το ίδιο θέμα για να αποφύγω να υπάρχουν προβλήματα ερμηνείας γιατί η νομική είναι πάντα σε θέση να εξετάσουν γιατί ο νομοθέτης εκείνο δικείμενο πήρε αυτή τη λέξη και στο άλλο κείμενο δεν πήρε την ίδια λέξη. Και έτσι ε, βασίζουν στον στην άμμο με μεγάλα νομικά επιχειρήματα, τα οποία όμως ε, σπέρνουν τη σύγχυση. Και τέλος, και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους να αντιδράσουν, τέλος θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι οι προτάσεις που γίνονται όσον αφορά τον καταθέτη στην έκθεσή μου είναι ισχυρότερες από εκείνες που εφαρμόζουν για τα OPCVM. Μου λέμε ότι εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Άλλο λόγο είναι πολύ απλός, δηλαδή τη στιγμή κατά την οποία η οδηγία για τα OPCVM παρουσιάστηκε, ήμασταν σε μία άλλη ε, σε ένα άλλο πλαίσιο και ελπίζω θα μπορέσει η δική μας ε, οδηγία να ε, διευρυνθεί για να καλύπτει τους καταθέτες και σε αυτή την οδηγία. Είναι νομικά δυνατό. Τελειώνοντας. Διάβασα μάλιστα ένα σχόλιο σε μια γαλλική κατηθετες και σε αυτη την οδηγια ειναι νομικα δυνατο τελειωνοντας διαβασα μαλιστα ενα σχολιο σε μια γαλλικη εφημεριδα που έλεγε ε, πολύ κακό για το τίποτα. Πρόκειται για το τίποτα όμως σε αυτή την πρώτη οδηγία. Δεν νομίζω. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε αρκετά ρεαλιστές για να λάβουμε υπόψη μας τις πτυχές που οικονομικά είναι χρήσιμες. Σημαίνει γιατί δεν θα πρέπει νομίζω να ευνοήσουμε, μάλλον θα πρέπει να εντεχθούμε στην πραγματική και καθαρή κερδοσκοπία. Από την άλλη μεριά κάθε φορά που αυτές οι οικονομικές δραστηριότητες έχουν ένα ε, όφελος οικονομικό δεν θα πρέπει να πλήξουμε την ανταγωνιστικότητα της ε, ευρωπαϊκής επικράτειας, αλλά θα πρέπει βέβαια να επαγρυπνούμε. Εκείνοι που νομίζουν ότι η κρίση ξεπεράστηκε γιατί οι τράπεζες βρίσκονται σε καλή υγεία και δίνουν πολλά, πολύ καλές πληρωμές. Ε, θα πρέπει να δούμε τι έγινε στις πρόσφατες μέρες στο Ντουμπάι. Και γι' αυτό θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Ε, θα πρέπει να προσθέσω ότι υπάρχουν ειδικέ περιπτώσεις που θα πρέπει να τι εξετάσουμε στενά, holding, investment trust, ε, κρυστά ταμεία στην Γερμανία. Θα πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς για να ξέρουμε κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί που είναι κάπως ιδιάζοντες θα πρέπει να ε, ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής οδηγίας. Τελειώντας, έχω να πω ότι η αρχή, σύμφωνα με την οποία κανένας τομέας των χρηματοπιστωτικών επαγγελμάτων δεν πρέπει να ξεφεύγει, αυτή θα είναι η αρχή που θα πρέπει να μας διέπει στις προσπαθίες μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ωραία πέρασε ο χρόνος μας ακούγοντας όλα αυτά που μας είπατε. Στην περίπτωση που κάποιον δεν είπα, μπορεί βεβαίως να ζητήσει το λόγο, θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές και μετά τους σκιώδεις θα μιλήσουν. Peter Skinner, Cool, uh, was somebody Μήπως ξέχασα κάποιον, κάποιος που δεν άκουσε το όνομά του. Okay, so, uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε και μόνο το γεγονός ε, ότι τόσοι πολλοί ζήτησαν το λόγο ε, διαψεύδει το γεγονός αυτό αυτά που αναφέρει στο γαλλικό τύπο ότι πολύ κακό για το τίποτα. Γιατί αν ήταν πολύ κακό για το τίποτα δεν θα ζητάγαν και τόσοι πολλοί το λόγο. Ζωάν Πόλ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που κατέθεσε στην, ε, το σχέδιο της έκθεσης. Επίτρεψε μου να σου παρουσιάσω την άποψη του σκιώδου συζητητού μας, του κ. Γκέμπελς, ο οποίος παρακολουθεί το θέμα εκ του σύνεγγης, αλλά αυτή τη βδομάδα δυστυχώς έπρεπε να ε, πάει ε, στη συνάντηση με τις χώρες ΑΚΕ, γιατί είναι και εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν λοιπόν κάποια σημεία τα οποία τα βρίσκουμε πάρα πολύ καλά στο σχέδιο της έκθεσης και όπου με απόλυτη σαφήνεια λέμε ότι ο Ζαν Πολ προχωράει περισσότερο και κάνει πολύ πιο καλές προτάσεις από ότι η Σουηδική Προεδρία. Παραδείγματο χάρη, αυτό ισχύει για τους τομείς εκείνους όπου ο στόχος είναι η έκθεση αυτή να συνδέει συνδεθεί με τη νέα Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, να δημιουργηθεί μια γέφυρα με άλλα εργαλεία όπως είναι η USITS και η MIFID. Το ίδιο ισχύει και για την διαγραφή των ε, ορίων, κάτι το οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό. Κατά την άποψή μας είναι σωστό το ότι το ευρωπαϊκό διαβατήριο, όπως λέγεται, που θα εκδοθεί, ε, το διαβατήριο αυτό θα προβλέπεται για τους ε, διαχειριστές που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα καλό ευρωπαϊκό ποιοτικό προϊόν. Εμείς ε, συμφωνούμε με την άποψη ότι πρέπει οι ε, οργανισμοί αξιολόγησης όχι μόνο να είναι ανεξάρτητη αλλά και το ότι τα κεφάλαια των ταμείων ε, θα πρέπει να αξιολογούνται διαφορετικά από τους μάνατζερ, από τους διαχειριστές. Θεωρούμε επίσης ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα προγράμματα ε, αποζημίωσης και αντιστάθμισης. Το ίδιο ισχύει και για τα κέρδη που θεωρούνται υπερβολικά. Ως εκ τούτου και αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό το πλαίσιο ε, και δεν θα πρέπει να την χάνουν ειδική σε φορολογικής μεταχείρισης. Όμως υπάρχουν και κάποια σημεία που θέλουμε να ασκήσουμε κριτική, όπου επιθυμούμε πιο ε, αποτελεσματικούς κανόνες. Παραδείγματο χάρη αυτό ισχύει για τη μόχλευση. Όλοι μιλάνε για τη μόχλευση, αλλά σε τελική ανάλυση δεν είναι δυνατόν οι ίδιοι οι διαχειριστές να αποφασίζουν πού θα περικοπεί η μόχλευσή τους, πού θα βρει τα όρια η μόχλευση. Εμείς πρέπει να τα ρυθμίσουμε αυτά. Και γι' αυτό λοιπόν ως πολιτική ομάδα εμείς θα τοποθετηθούμε επί του θέματος για να σας πούμε τι ακριβώς ε, πιστεύουμε. Κατά τα άλλα, ε, επιθυμούμε να απαγορεύονται ε, ζημιογόνες ε, συναλλαγές του αέρα. Επίσης, το empty voting ή οι μυστικές αγοραπολισίες και αυτά πρέπει να ρυθμίζονται γιατί και εδώ θεωρούμε ότι ελοχεύουν κίνδυνοι. Το ίδιο ισχύει και για τα asset stripping. Αυτό το βρίσκουμε ζημιογόνο για πολλές επιχειρήσεις αν τελικά δεν βρούμε νέες μορφές κανονισμών. Εν κατακλείδη λοιπόν, θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν πάρα πολλά για την έκθεση και πέρα από το σχέδιο, κυρίως όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τις πληροφορίες, κυρίως προς όφελος των ε, ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές. Σε τελική ανάλυση δεν θα κατορθώσουμε να επιζήσουμε αν δεν υπάρξει ένας σαφής ορισμός των ελάχιστων ιδίων κεφαλαίων που είναι απαραίτητα για τα επενδυτικά ταμεία. Κυρίες και κύριοι, η κρίση έφερε όλους μας σε μια κατάσταση όπου επιτέλους, και το υπογραμμίζω επιτέλους, θα κατατεθούν νομοθετικές προτάσεις. Εδώ λοιπόν καλούμεθα να δραστηριοποιηθούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ υπογραμμίζω ότι ο Ζαμπόλ δικαίως είπε ότι δεν πρέπει να παραμείνει κανένα επικίνδυνο προϊόν αρρύθμιστο. Αυτό ισχύει όχι μόνο για την ενεργό πλευρά της πρόθεσης προϊόντων, αλλά και για την παθητική. Εμείς λοιπόν εδώ θα στηρίξουμε ενεργά τον εισηγητή και βεβαίω θα καταθέσουμε και τις δικές μας τις συμπληρωματικές προτάσεις. Ο κύριος Κρέντς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας, τον Ζαν Πολ Γκουζές, γιατί πραγματικά προσπάθησε με εκατοντάδες ε, τροπολογιών παρόλα αυτά να προχωρήσει την πρότασή του. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες θα ε, επηρεαστούν, θα θυχτούν από αυτή την ε, οδηγία εγώ εξακολουθώ να έχω αμφιβολίες κανονικά θα έπρεπε να ασχοληθούμε περισσότερο με τα hedge funds και με τα ιδιωτικά κεφάλαια επενδύσεων αλλά τι έγινε τελικά μπήκαν εκεί πέρα όλα όσα ε, δεν είναι usage αυτά τα αυτοδιαχειριζόμενα κεφάλαια όπως είναι παραδείγματος χάρη τα χρηματιστήρια στη Μεγάλη Βρετανία ή τα επενδυτικά ταμεία που υπάρχουν στην Σουηδία ή τα ειδικά επενδυτικά κεφάλαια που υπάρχουν στη Γερμανία, αυτά δεν αποτελούν συστημικό κίνδυνο. Αυτά έτσι και αλλιώ ε, ρυθμίζονται και υποπτεύονται παρκώ. Καμία δουλειά δεν έχουν αυτά εδώ μέσα. Να φύγουν, να εξαιρεθούν. Γι' αυτό λοιπόν, όσον αφορά το πεδίο τη εφαρμογή, να, ήδη σα έκανα κάποιε παρατηρήσει. Κατά τα άλλα, συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφο κ. Μπούμαν, ότι ο Ζαν Πολ ε, παρουσιάζει μια σειρά από πολύ καλές ε, θετικές προσεγγίσεις, όμως εγώ έχω να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Πρώτον, συμφωνώ ότι πρέπει να καταργήσουμε το κατόφλι. 100 εκατομμύρια ή κάποιο άλλο ποσό που αναφέρεται. Αυτά όλα τι είναι, δεν λένε τίποτα. Άντε να είναι 57 και όχι 58. Καμία σχέση δεν έχουν όλα αυτά. Να μην υπάρχει κατόφλι. Όμως παρόλα αυτά θεωρώ ότι θα έχουμε πολλή δουλειά αν ασχοληθούμε με το θέμα της αναλογικότητας που προσέθεσε ο Ζαν Πολ. Αν θέλουμε να του δώσουμε σάρκα και οστά. Όσον αφορά τώρα τις ε, τρίτες χώρες, πράγματι αυτό δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, διότι κατά τη δική μου την άποψη την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να την αποκλείσουμε από τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ευρώπη δεν πρέπει να γίνει ούτε οχυρό ούτε σοφρονιστικό κατάστημα. Είναι λοιπόν σημαντικό ε, το τι λύση θα αναζητήσουμε. Ε, πρέπει να σας πω, συμφωνώ ότι το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο θα πρέπει να χορηγείται μόνο σε ένα διαχειριστή ο οποίος έχει την έδρα του στην Ευρώπη και το ίδιο ισχύει και για το επενδυτικό ταμείο το οποίο διαχειρίζεται. Στην περίπτωση αυτή συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να παραμένει ανοιχτή δυνατότητα για τους Ευρωπαίους επενδυτές να επενδύουν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ εγώ έχω κάποιο πρόβλημα. Εσύ λες, ναι εντάξει αυτό γίνεται με βάση ε, τα καθεστώτα που υπάρχουν ε, τα μεμονωμένα 27 στα 27 κράτη-μέλη υπό την προϋπόθεση ότι κάθε μία από αυτές τις χώρες, άρα δηλαδή 27, κάθε μία από αυτές θα πρέπει να συνάψει μία διμερή συμφωνία με τη χώρα στην οποία έχει την έδρα του το Ταμείο. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ περίπλοκο και τελικά θα οδηγήσει στο ότι ε, θα πρέπει ένα κράτος όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες παραδείγματο χάρη να ε, υποβάλει 27 διαφορετικές αποδείξεις. Αυτό κατά πόσο είναι εφικτό το αμφισβητώ. Όσον αφορά τώρα τις ε, τράπεζες παρακαταθήκης. Αναφέρθηκε από τον Ζαν Πολ ότι αυτές οι τράπεζες παρακαταθήκων πρέπει να ε, ρυθμιστούν μαζί με τα κανονικά επενδυτικά ταμεία ή κεφάλαια. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε την πρόταση της Κομισιόν. Η Κομισιόν ε, πρόκειται να ρυθμίσει αυτές τις ε, τράπεζες παρακατευτικών, να εκπονήσει ρυθμιστικούς κανονισμούς και σε τελική ανάλυση θα πρέπει να προκύψει κάτι που να είναι λογικό. Δηλαδή οι απαιτήσει απέναντι σε μια τράπεζα παρακαταθήκων η οποία αυτή τη στιγμή λειτουργεί για τις εναλλακτικές επενδύσεις και η οποία κατ' ουσίαν λειτουργεί και για τους θεσμικούς επενδυτές, αυτές οι τράπεζες δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μεγαλύτερες επενδύσεις από τα, τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα επενδυτικά ταμεία. Ίσως ε, ε, θα πρέπει οι ρυθμίσεις να είναι ε, περισσότερο αυστηρές στα usage και όχι τόσο στους εναλλακτικούς επενδυτές. Όσον αφορά την ανεξαρτησία των οργανισμών αξιολόγησης, των αξιολογητών. Συμφωνώ απόλυτα. Ο καθένας μπορεί να πει αν έχει ανεξάρτητο αξιολογητή ή όχι και εγώ συμφωνώ. Ε, βασικά πρέπει να σας πω ότι είμαι κατά αυτού του θεσμού γιατί αυτός ο φερόμενος ε, ανεξάρτητος ε, εκτιμητής είναι όπως αυτη οι περίφημοι οργανισμοί αξιολόγησης. Κατ' ουσίαν δημιουργούμε και πάλι ένα μονοπόλιο προστίθενται οι δαπάνε. Εγώ εξακολουθώ να έχω εδώ τι επιφυλάξει. μου και έρχομαι σε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Σε τελική ανάλυση όταν ε, ή αν θελήσουμε να εισάγουμε μια τέτοια οδηγία πρέπει να διερωτηθούμε ποιο είναι ο στόχο μα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πεπισμένοι ότι εισάγοντα αυτή την οδηγία πράγματι κάτι θα αλλάξουμε. Μέχρι τώρα είχαμε εμβαλωματικές ε, αλλαγές και βελτιώσεις αλλά δεν είχαμε ριζική αλλαγή αυτές οι εταιρείε που αναφέρονται, είτε είναι ιδιωτικών κεφαλαίων, είτε είναι hedge funds, κατ' ουσίαν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν όπως μέχρι τούδε. Και ε, την πρακτική θα μπορέσουμε να την αλλάξουμε μόνο αν επέμβουμε στη μόχλευση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές το τι ακριβώς κάνουμε και ποια είναι η στάση μας απέναντι στα ίδια κεφάλαια. Να πούμε 120 ή 130 χιλιάδες ε, ελάχιστο ε, κεφάλαιο ελάχιστο ποσό ιδίων κεφαλαίων για μια επενδυτική τράπεζα Πώς ασχολούνται με επενδύσεις, όπως είπε και μια ελβετική τράπεζα. Ε, αν, παραδείγματο χάρη, ένα ε, ταμείο είναι μέρος μιας τράπεζας, θα πρέπει και αυτό να έχει ίδια κεφάλαια όπως και η τράπεζα. Αν χρηματοδοτείται από την τράπεζα, τότε η χρηματοδότηση του Ταμείου από την Τράπεζα θα πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο το επιτόκιο θα πρέπει να καλύπτει και τους κινδύνους. Άρα δηλαδή από το ύψος του επιτοκίου θα μπορούμε να κατανοούμε κατά πόσον το Ταμείο κινεί μεγάλα ποσά ή όχι. Και τέλος θα πρέπει να σκεφτούμε πώς ακριβώς θα περιορίσουμε τη μόχλευση. Και αυτό δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών. Νομίζω ο Ζαν Πολ εδώ είσαι πολύ καλόπιστος. Ε, ο ένας διαχειριστής ε, κεφαλαίων, κάποιος ε, μπορεί να έχει συνηθίσει να τρέχει με την πέμπτη ταχύτητα, να επενδύει με ταχύτητα, να, να κάνει κινήσεις πάρα πολύ γρήγορες. Άλλοι διαχειριστές πάλι είναι πιο συντηρητικοί. Η εποπτεία θα πρέπει να γίνεται μέσα από τις εποπτικές αρχές. Και άλλα δύο σημεία. Στην περίπτωση αυτή συμφωνώ με τον Ούντο ότι ε, τουλάχιστον θα πρέπει να απαγορεύσουμε τις συσσαγωγικά γυμνές αγοραπολισίες. Γυμνές αγοραπολισίες κατά την άποψή μου είναι απόλυτα αρνητικές. Εγώ δεν κατανοώ πώς μπορούμε να επιτρέψουμε σε κάποιον με τέτοιου είδους αγοραπολισίες να επηρεάζει καθοριστικά μία αγορά. Αυτό είναι ρουλέτα. Ρουλέτα εις βάρος κάποιων που δεν συμμετέχουν, που είναι απλοί επενδυτές και των οποίων όμως οι μετοχές ξαφνικά ακολουθούν μια κατεύθυνση που δεν μπορούσαν καν να φανταστούν. Ε, short selling, ναι, αλλά naked short selling επουδενή. Και ε, τέλος, ε, Jean αυτά που λες στο σημείο 13 Καλά και σωστά είναι αυτά, πράγματι προσπάθησε και εσύ και εμείς οφείλουμε να μεριμνήσουμε αυτή ε, η, το σχέδιο ρύθμισης που βρίσκεται κάτω από πίεση να μην βρεθεί σε αντίφαση με άλλα σχέδια τα οποία επεξεργαζόμαστε. Να συμφωνήσουν αυτά με το usage, με το MIFID, ε, με όλα αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και κατά τα άλλα συμφωνώ μαζί σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή μου. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά του. Ήταν πολύ ανοιχτός, έτεινε ευήκον ους, είπε θα ακούσω, άκουσε. Είπε θα γράψω, έγραψε. Ελπίζω στο επόμενο στάδιο να πει θα δεχτώ και κάποιες από τις τροπολογίες σου. Αναγνωρίζει και άλλες οντότητες πέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο χαιρετίζουμε και αναγνωρίζει και τις υφιστάμενες πρακτικές. Αναφέρει ας πούμε τους prime brokers. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς αυτό που μας νοιάζει είναι πώς αυτό το νομοθέτημα θα επηρεάσει τη ζωή των εργαζομένων, των συνταξιδοτών, των επενδυτών. Και πώς θα αποφύγουμε περί του κινδύνου. Και βεβαίω, να έχουμε ένα πλαίσιο εντό του οποίου οι συναλλασσόμενοι θα αισθάνονται και θα είναι ασφαλείς. Συμφωνώ με τον Ζων Πολ για το ότι αναφέρει τα εθνικά συστήματα τα συντοξιδοτικά εννοώ ότι δεν υπάρχει περιθώριο συντονισμού ή μάλλον εναρμόνισης. Είναι σημαντικό βεβαίω να μην περιπλακεί παραπάνω το σύστημα για τους επενδυτές στην Ένωση που θέλουν να συνεχίσουν να επενδύουν σε αυτά τα προϊόντα και αυτά τα ταμεία. Ιδιαίτερα τα ταμεία τα οποία συμμετέχουν σε αναπτυξιακά προγράμματα. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε επενδυτές από τον επενδύουν τα χρήματά τους σε τέτοιου προγράμματα. Επίση χαιρετίζω το γεγονό ότι η οδηγία αυτή είναι συνεπής με τις άλλες οδηγίες. Η συνέπεια είναι πολύ σημαντικό. και η εξολόγηση του τι είναι αναλογικό, του τι είναι λογικό. Μ' αρέσει. Αυτά είναι αυτά που με βρίσκουν σύμφωνο. Οι ανησυχίε μου τώρα. Το είπα και πριν για την ανάπτυξη και την, ε, τα αναπτυξιακά προγράμματα. Οι Ευρωπαίοι επενδυτές ...ως επενδύουν δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν τα χρήματά τους σε προγράμματα αναπτυξιακού περιεχομένου. Αυτό δεν είναι για να κάνουμε λιγότερο φτωχές στις αναπτυσσόμενες χώρες μόνο, είναι για να υπάρχει μια υγιής οικονομία. Για τις νήσους Κέιμαν είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που προσπάθησε να βγει από τη φτώχεια περνώντας κατευθείαν στις δημοσιονομικέ υπηρεσίες, χωρίς να περάσουν από τη γνωστή αλυσίδα γεωργία μικρή κλίμακο, γεωργία μεγάλης κλίμακο, βιομηχανία, υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό, θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούν μαζί μας. Ε, Μην με παρεξηγήσετε, έτσι. Δεν εννοώ ότι θα πρέπει να του δώσουμε λευκή επιταγή, και όντω πρέπει να ανυψώσουν τι προδιαγραφέ του και το πρότυπά του εάν θέλουμε να υπάρχει πλήρη συνεργασία. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έκαναν αυτή την προσπάθεια. Τώρα, για τα αποθετήρια και την προστασία των επενδυτών. Θέλω να είμαστε συνεπεί. Όλοι μα σε αυτή την Επιτροπή αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να διδαχθούμε από τα παρελθόντα σφάλματα. Δεν είναι δυνατόν να εγκρίνουμε νομοθεσία η οποία να μην λαμβάνει υπόψη τη να την ιστορία. Το θέμα του κινδύνου. Ξέρω ότι το έχουν ε, προωθήσει πολύ οι σοσιαλιστές. Και συμφωνώ. Αλλά υπάρχουν λόγοι για την αποτυχία. Οι Lehman Brothers. Οι Lehman Brothers χρησιμοποίησε αποθετήρια μεταξύ διαφόρων επενδυτικών ομίλων. Για να είμαστε συνεπείς, θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη δυνατότητα στους τραπεζικούς ομίλους να χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο. Δεν έχω καταλήξει σε α, μονοσήμαντη ερμηνεία ή απάντηση, αλλά ακόμα υπάρχουν επενδυτές που περιμένουν το μερισμά τους, που τους είπαν ε, ότι θα το πάρουν σε 10 χρόνια. Το αναφέρω ως ένα σημείο συζήτησης για το μέλλον. Ευχαριστώ, Ζων Πολ. Και είμαι στη διάθεση βεβαίω όλων και του εισηγητή και των ε, σχεδόν για να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Πασκάλ Κάμπερ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον Ζων Πολ Γκοζέθ που όντως έκανε πολύ ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική δουλειά με ανοιχτό πνεύμα με όλους τους σκιώδεις. Βεβαίω, δεν θα σα εκπλήξει ότι θα διαφωνήσω απόλυτα με τον συντηρητικό, Βρετανό συνάδελφο που μόλις μίλησε. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι τα επενδυτικά αυτά τα μία είναι ένα μέσο καταπολέμησης της στόχιας στον κόσμο και καλό πράγμα. Δεν το είχα σκεφτεί. Το ομολογώ. Πάντως εμείς ως πράσινοι υποστηρίζουμε το περιεχόμενο των εξελίξεων. Το πρώτο, η πρώτη εξέλιξη είναι μια συνολική προσέγγιση δηλαδή, χωρίς όρια και κατόφλια, αλλά με την αρχή της αναλογικότητας. Το δεύτερο στοιχείο είναι η ενσωμάτωση του θέματος των αμοιβών στο κείμενο αυτό, που απουσίαζε για λογικούς λόγους ο χρονοδιαγράμματος όταν η Κομισιόν έκανε το πρώτο σκαρίφημα της ε, οδηγίας είναι νομίζω αντικείμενο συνένεση να συμβληθεί το, το θέμα των αμοιβών στο κείμενο. Και βεβαίω το τρίτο είναι του ΕΣΜΑ ω ένα βασικό στοιχείο ρύθμιση των επενδυτικών ταμείων. Κάτι το οποίο και αυτό είχε αποκλειστεί από την αρχική εκδοχή της πρόταση της Κομισιόν. Τώρα, οι διαφωνίες μας ποιε είναι με την έκθεση αλλά και το σημείο ισορροπία αυτή. Πρώτα απ' όλα, ερμηνεύουμε την έκθεση με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ανέφερε ο κύριος Κέντς ότι εμποδίζουμε τους Ευρωπαίους επενδυτές να επενδύσουν σε ταμεία εκτός Ένωσης και ότι αναδιπλωνόμαστε στα πλαίσια της λογικής της Ευρώπης οχυρού. Όχι. Εμείς έχουμε την εντυπωσία ότι αυτή η έκθεση ανοίγει διάπλατα την πόρτα στη δυνατότητα οι Ευρωπαίοι επενδυτές να βάλουν τα χρήματά τους σε επενδυτικά ταμεία τα οποία ε, τα διαχειρίζονται κάποιοι εκτός της Ένωσης. Διότι η μόνη προϋπόθεση που αναφέρεται για να μπορεί κανείς να επενδύσει σε τέτοιου είδους εναλλακτικά ταμεία εκτός Ένωσης είναι ο σεβασμός και μόνο των διεθνών προτύπων. Διεθνά πρότυπα, γιούσκο δηλαδή. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά αν είναι έτσι τα πράγματα, αυτό σημαίνει ότι μόνο τα πρότυπα γιούσκο επιβάλλουμε, επί των οποίων δεν υπάρχει καμία συμφωνία για το πώς θα εφαρμοστούν από τους επόπτες. Δηλαδή υπάρχει μια θεωρητική συμφωνία αλλά δεν υπάρχει καμία συμφωνία για το πώς ελέγχουμε την εφαρμογή αυτών των προτύπων. Είναι λοιπόν θεωρητικά μόνο πρότυπα και καθόλου πρακτικά. Γι' αυτό και ακριβώ το λόγο, ο επόπτης από τι νήσου Κέιμαν προσυπέγραψε τα πρότυπα αυτά, διότι ιδάλω δεν θα τα προσυπέγραφε ποτέ. Γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτή η θέση είναι πιο χαλαρή εναντί τη αρχική θέση τη Κομισιόν, που ήταν πιο στεναρή. Ένα ελάχιστο τουλάχιστον πρότεινε, το οποίο εξαφανίστηκε τώρα, δηλαδή την υπογραφή μια συμφωνία συνεργασία στα φορολογικά θέματα επί τη βάση των προτύπων του ΟΣΑ. Δηλαδή δεν υπάρχουν μόνο τα εκ των πραγμάτων πρότυπα τη Ιούσκο που είναι εντελώ μινεμαλιστικά αλλά υπάρχει τουλάχιστον μια συμφωνία για τα φορολογικά πρότυπα του ΟΣΑ που δεν μα καλύπτουν, συμφωνούμε, αλλά που είναι αν μη τι άλλο ένα το κρατούμενο. Είναι παράδοξο λοιπόν να μιλάμε για αυτό με την ανταλλαγή πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην λαμβάνουμε καθόλου υπόψη αυτό όταν συζητούμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Κάτι άλλο με το οποίο διαφωνούμε. Είναι η μοχ, ο μοχλός, η μόχλευση. Στην αρχική πρόταση της Κομισιόν προβλεπόταν η δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να ελέγχει τη μόχλευση και τα κράτη-μέλη σε εξαιρετικές περιπτώσεις να μπορούν να επιβάλλουν και άλλες εξαιρετικές εξαιρετικούς περιορισμούς. Αυτός ο μόνιμος έλεγχος δεν υπάρχει πια και μιλάμε μόνο για απλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του διαχειριστή και της ΕΣΜΑ. Και η έκθεση, στην τροπολογία υπερθμών 100 δεν απατώμε, λέει ότι η ΕΣΜΑ μετά αποφασίζει αν ο μοχλός ε, είναι ε, πολύ υψηλό, στην περίπτωση στην οποία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εκτός από εξαιρετικέ περιστάσεις, λέει η έκθεση. Εκεί, εντάξει, μπορούμε να δράσουμε, όπως προτείνει η Κομισιόν. Οι εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι δεν είναι δυνατόν να δράσουμε μόνο σε εξαιρετικέ περιστάσει για να περιορίσουμε το μοχλό. Όχι. Πρέπει να το προλάβουμε. Πρέπει εξάντε να έχουμε τη δυνατότητα είτε μέσω της ΕΣΜΑ είτε μέσω άλλου φορέα να ελέγχουμε το μοχλό. Και βεβαίως ακόμα περισσότερο στις εξαιρετικές περιστάσεις. Πρέπει να αντιστρέψουμε λοιπόν τη λογική που διέπει την έκθεση αυτή για να συνάδουμε περισσότερο με την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω, διότι δεν σημαίνει και καθημερινά οι πράσινοι να υποστηρίζουν πρόταση της Κομισιόν. Έτσι. Επίσης κάτι σημαντικό είναι ο ρόλος της ΕΣΜΑ. Ο ρόλος της ΕΣΜΑ σε σχέση βεβαίω με την οδηγία για την ε, εποπτεία. Αλλά αν δημιουργήσουμε ευρωπαϊκή αγορά αν δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο θα έπρεπε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή διαπίστευση και ένας φορέας μόνο διαπίστευση των ταμείων εκείνων που θα ζητούν τη βούλα, τη σφραγίδα την ευρωπαϊκή. Αυτό για να αποφευθούν συγκρούσει ερμηνεία ε, και αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορών, διαφορετικών εθνικών ε, εποπτικών οργάνων. Το τελευταίο μου σχόλιο αφορά την αρχιτεκτονική ή αν θέλετε τη δυναμική αυτού του κειμένου. Δημιουργούμε ουσιαστικά δύο αγορές. Μία αγορά με ευρωπαϊκό διαβατήριο που περιορίζεται στα ταμεία τα οποία διαχειριζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά όλα τα υπόλοιπα με διαφορετικό καθεστώς και τη δυνατότητα οι τρίτες χώρες να θέτουν ε, σε κυκλοφορία χωρίς πολλούς περιορισμούς τα ταμεία τους ε, που ε, έχουν έδρα τρίτες χώρες εκτός Ένωσης η χρηματοοικονομική ροή θα στραφεί προς ένα ρυθμισμένο περιβάλλον, το ευρωπαϊκό, με το ευρωπαϊκό διαβατήριο κτλ. Ή μήπω θα πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή στα ταμεία που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι το μέγα στίχημα. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι επί της αρχής να το αναλάβουμε αυτό το στίχημα αυτή την πρόκληση, αλλά έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι τα ταμεία έχουν κάθε όφελος να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο για την προστασία των επενδυτών, αλλά και για το City, δηλαδή τη Βρετανική χρηματαγορά. Και φαντάζομαι θα συμφωνεί ο Βρετανός συνάδελφος με αυτό που λέω. Το σημείο ισορροπίας του κειμένου δεν είναι τελικά, δεν μπορεί να είναι μια ενθάρρυνση στα επενδυτικά αυτά τα μία να φύγουν από την Ένωση και να πάνε σε τρίτες χώρες. Έτσι όπως είμαστε με αυτό το διτό καθεστώς, τα πράγματα νομίζω ότι είναι καλύτερα. Δηλαδή θα έχουμε στοιχεία που θα προστατεύουν και τους επενδυτές στην Ευρώπη, αλλά και την πίσνα στο City. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον Ζαν Πολ. Νομίζω ότι έκανε πάρα πολύ δουλειά. Το βλέπει κανείς αυτό, ακόμα και αν διαφωνεί μαζί του. Αλλά τουλάχιστον ε, πραγματικά ασχολήθηκε σε βάθος με το θέμα και γι' αυτό τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την άποψη της, ε, των αριστερών, της ΓΚΟΕ, θέλω να πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό για μας. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε όλα τα ταμεία. Αυτό είναι απόλυτα σαφές. Ε, είναι σαφές και αυτονόητο, αλλά εγώ ήθελα να το πω. Υπάρχουν ε, και άλλες δυνατότητες και άλλοι τρόποι να αποκτήσει η οικονομία κονδύλια. Δεν είναι μόνο τα hedge, fund, hedge funds. Αυτά τα hedge funds ε, έχουν, επηρεάζουν την αγορά εργασίας, τα ταμεία, τα ασφαλιστικά, την ανεργία και αυτό δεν είναι καλό και το λέω ευθύ εξ αρχή. Γνωρίζω βέβαια ότι μπορούμε να συζητήσουμε περαιτέρω για το κατά πόσον η οδηγία αυτή ε, μπορεί να παρεμποδιστεί ή όχι. Κατά τη δική μου άποψη και τη δική μας, αυτό που είναι ιδιαίτερα ευχαριστώ, ευχάριστο είναι ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ρύθμιση. Εμάς ως αριστερά μας ε, ενδιαφέρει, αν δεν μπορούμε να αποφύγουμε την αγορά, τουλάχιστον να τη ρυθμίσουμε όσο περισσότερο γίνεται η δουλειά του Ζαν Πολ ε, τουλάχιστον ε, δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ρύθμιση. Αυτό το χαιρετίζουμε. Το να διαγραφούν ε, τα όρια, το κατόφλι, αυτό και εμείς το βρίσκουμε σημαντικό. Τώρα, αυτά που λέξαν για τη μόχλεψη, εγώ δεν θέλω να τα επαναλάβω νομίζω ότι όπως τα καταλάβαμε και όπως τα επενήχθη ο μιλητής, εμείς τα στηρίζουμε. Μπορούμε να φανταστούμε ότι τέτοιου δυνατότητες θα πρέπει να απογορευθούν πλήρως. Και βεβαίως αυτό ε, θα το επιδιώξουμε μέσα από τροπολογίες. Ε, το naked short selling, αυτό είναι κάτι ε, το οποίο θα μας άρεσε να απογορευθεί. Ε, σας είπα, αν τελικά περάσει η οδηγία, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Και κάτι άλλο, ε, τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εγώ χθε συμμετείχα σε μία συζήτηση στην Αυστρία, όπου συζητήθηκε και εκεί το θέμα. Το θέμα του δικαιώματος ε, συναπόφασης, ε, η συμμετοχή των συνδικάτων σε επιχειρήσεις ε, που επηρεάζονται από επενδύσεις. Αυτό εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα θελήσουμε πραγματικά να εκπονηθούν οι κανισμοί εκείνοι που ε, θα επιτρέπουν μεγαλύτερη δυνατότητα συναπόφασης από ό,τι μέχρι τώρα. Ε, κατά τα άλλα δεν θέλω να πω τίποτα άλλο γιατί τα περισσότερα που θέλω να πω ήδη ελέγχθησαν. Καλώς. Έχουμε μακρύ κατάλογο ομιλητών και όπως είπαν οι σκιώδεις δεν υπάρχει χρόνος, οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να περιοριστείτε σε δύο λεπτά της ώρας. Ο κάθε ομιλητής να έχει δύο λεπτά της ώρας, τόσο ώστε να έχουμε κάποιο χρόνο μετά για την Κομισιόν και τον εισηγητή. Η κυρία Φόρντ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ γρήγορη. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικό έργο του κυρίου Γκόζες. Καθόλου δύσκολο. Έβγε Και αυτό που μας ενδιαφέρει πιστεύω είναι η πραγματική οικονομία. Πώς επηρεάζουν αυτές οι οδηγίες, τις αναφιόμενες αγορές, τα συνταξιωτικά ταμεία και τα μυρίσματα αυτών, τα κεφάλαια κινδύνου, που είναι πολύ σημαντικά για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, για τις αναφιόμενες, για τις αναδιόμενες αγορές. Η ευθύνη του αποθετηρίου μπορεί να είναι μεγάλη τροχοπέδη για τις επενδύσεις στις αναδυόμενες αγορές. Και θα πρέπει να κινηθούμε σύμφωνα με την τροπολογία 79 για τις επενδύσεις στα, στα εξωτερικά ταμεία. Είχα θέσει ένα ερώτημα. Η εναλλακτική πόσο θα κόστιζε 15 με 20% του συνολικού μου εισοδήματος αν είμαι συνταξιούχος, τεράστιο ποσό. Χαίρομαι λοιπόν που διευκολύνουμε τους Ευρωπαίους επενδυτές να συνεχίσουν να επενδύουν εκτός Ένωσης. Πάντως με ανησυχεί η τροπολογία 17. Οι ιδιωτικές συντάξεις δεν ξέρουμε πώς ακριβώς έχουν προς το παρόν αν θα πρέπει να στραφεί κανείς πάλι στον ρυθμιστή στη χώρα καταγωγής για να δούμε αν συμφωνεί. Αν είναι δηλαδή ένα hedge fund το αμερικανικό, το SEC θα πρέπει να έχει συμφωνία με 27 διαφορετικά κρατημέλη. Αυτό μου φαίνεται κάπως έτσι ότι χωλαίνει ως λύση. Αφήστε δε που θα έχει και πολύ σημαντικές επιπτώσεις στη σύνταξή μου για τα κεφάλαια κινδύνου, για τα επενδυτικά κεφάλαια κινδύνου. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε δυσκολίες με αυτή τη νέα πρόταση. Για τα αποθετήρια επίσης, επειδή υπάρχουν τόσο λίγα, μπορούμε να δημιουργήσουμε, μπορεί να δημιουργήσουμε ένα συστημικό κίνδυνο με τη μείωσή τους. λέμε το απευθυντήριο θα πρέπει να είναι στο ίδιο κράτο μέλο με το ταμείο. Θα πρέπει να το δοκιμάσουμε αυτό ως λύση. Αν το δέχεται και ο κλάδος, αν είναι αποτελεσματικό. Και κάτι τελευταίο για την ΕΣΜΑ. Ανησυχώ, γιατί εκχωρούμε πολλέ αρμοδιότητες που δεν έχουν ακόμα συζητηθεί και συμφωνηθεί. Η ΣΥΖΑΡ αποτελείται από 30 ανθρώπους. Τώρα θα είναι 80 στην ΕΣΜΑ. Η FSA έχει 3.000 ανθρώπους προσωπικό. Δεν τα έκανε και όλα τέλεια η FSA, έτσι. Η ΕΣΜΑ θα βρει τους σωστούς ανθρώπους. Για το μοχλό, ομιλώ. Ή μήπως θα πρέπει να τα διαχειρίζονται όλα αυτά οι εθνικές αρχές και μετά η ΕΣΜΑ να βάζει το τελικό φρένο. Η κυρία Λούλινγκ χωρίς μικρόφωνο δεν την ακούμε. Με μικρόφωνο την ακούμε. Θα ξαναρχίσω από την αρχή γιατί θέλει ο κύριο Γκοζέ να καταλαβαίνει τι λέω. Από τη μετάφραση. Αστείευεται η κυρία Λόλινγκ εφόσον μιλάει γαλλικά. Δηλαδή την ίδια γλώσσα με τον κύριο εισηγητή. Ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί είναι ανοιχτός σε εξέβρεση ισορροπίας. Θα υποστηριχθεί το κείμενο από μεγάλη πλειοψηφία. Και εγώ διάβασα τον τύπο, τον γαλλικό κυρίως. Όντως, αναφέρονται πολλές κριτικές και επικρίσεις. Αλλά η γενική προσέγγιση, ο γενικός προσανατολισμός της έκθεσης εφόσον δεν αρνείται κάθε ρύθμιση, εφόσον δεν πρεσβεύει αυτό, είναι μια καλή βάση εργασίας. Και επειδή είσαι πολύ καλός διαπραγματευτής, Ζων Πολ, κατάφερες, δεν λέω να τετραγωνίσεις τον κύκλο, αλλά τέλος πάντων να τα πεις με τρόπο που βρίσκει τους περισσότερους σύμφωνους. Είμαι ικανοποιημένη λοιπόν. Και είναι πολύ σωστό και δικαιολογημένο το γεγονός ότι συμπεριέλαβε και τα κεφάλαια κινδύνου είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για τα ταμεία των τρίτων χωρών, που είναι το πιο επίμαχο κατά την άποψή μου θέμα και το πιο περίπλοκο θα πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένα πράγματα. Οι διατάξει για τα ταμεία των τρίτων χωρών και τι ε, συνθήκε κατανομή του, διανομή του μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζω ότι είναι σαφεί. Σύμφωνα με το σχέδιο έκθεση, τα ταμεία των τρίτων χωρών μπορούν να διανέμονται ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των καθεστώτων ε, επενδύσεων των ιδιωτικών εθνικών καθεστώτων, χωρίς να σέβονται αναγκαστικά τα ελάχιστα πρότυπα. Αυτό θα δημιουργήσει στρέβλωση, διότι στην αγορά μια ίδια χώρα θα έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ δύο ειδών ταμείων. Αυτά που ρυθμίζονται και αυτά που δεν ρυθμίζονται. Τα μία που θα εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Διαβατήριο, είτε του συγκεκριμένου κράτου μέλου είτε άλλων κρατών μέλων, μελών, και από την άλλη τα ταμεία των τρίτων χωρών που δεν θα καλούνται να σέβονται την οδηγία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρα συγκριτικό πλεονέκτημα, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ως εκ τούτου στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ενώ εμείς θέλουμε ισότιμη μεταχείριση. Η τροπολογία 62 προβλέπει ότι ο καταθέτης από κοινού με την εταιρεία διαχείρισης των περισσιακών στοιχείων υπολογίζει την καθαρή άξια και ζητώ να μου πείτε ποιο είναι το νόημα αυτής της τροπολογίας σε περίπτωση προβλήματος. Δεν θα ήταν πιο εύκολο μία οντότης να είναι υπεύθυνη και για τις δύο αυτές πτυχές. Αντί να αναφέρουμε ότι υπάρχει ευθύνη και από δύο οντότητες. Εγώ αυτό πιστεύω ότι περιπλέκει τα πράγματα για τον επενδυτή. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Είπε μου, έχω εμπιστοσύνη στον εισηγητή. Έχει πολλή δουλειά ακόμα βέβαιως να κάνει και δεν έχει οριμάσει να βγει από το πιεστήριο αμέσως. Ευχαριστώ. Θα επιταχύνουμε κάπως. Ευχαριστώ που το είπατε. Να επιταχύνουμε που μου δώσετε με τον λόγο. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το πολύ εντυπωσιακό του έργο που τονίζει όλα τα κύρια θέματα γιατί ενοχλήθηκα που κι άλλοι τον συνεχάρισαν. Αυτό οφείλεται όμως στην ε, ρεαλιστική προσέγγιση του εισηγητή που τονίζει τα σημαντικά θέματα και αυτό μας βοηθάει να συνεργαστούμε για το θέμα. Αυτό που είδαμε στην κρίση ήταν η έλλειψη διαφάνειας και η έλλειψη διακανονισμού. Θα πρέπει να είναι συνεπής με την πραγματική εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών αγορών τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό είναι το κύριο μενέκτημα και τώρα όταν προχωρήσουμε θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ταυτόχρονα να δώσουμε μακροπρόθεσμα στην οικονομική ανάπτυξη σταθερότητα. Γιατί κοιτάξτε, ο κύριος μας ε, στόχος είναι να ε, είμαστε ασφαλείς για να έχουμε περισσότερες επενδύσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Εύρος της οδηγίας. Θα πρέπει να εξετάσουμε ποιες είναι οι διαφορετικές δυνατότητες. Εμείς, εγώ δεν θέλω να καταλέξουμε σε μια κατάσταση στην οποία ε, προωθούνται τα εναλλακτικέ επίσης Έριξον. Οι σήμε δεν θα πρέπει να τύχουν αυτή τη αντιμετώπιση και θέλω να ρωτήσω τον εισηγητή, δεν θα μπορούσε να μελετήσει κατά πόσον. Όχι να κάνουμε μια εξαίρεση για κάποια επιχειρήση, αλλά για εταιρείε παραδείγματο χάρη που ε, ε, είναι στα, έχουν μπει στο χρηματοστήριο. πρέπει εδώ να ε, θεωρηθούν εναλλακτικά ε, συστήματα επενδύσεων. Και θα μπορούμε να προσθέσουμε ότι δεν πρόκειται να κερδίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν εξαιρέσουμε ε, αυτούς από τον, τα μέλη του κόσμου που έχουμε τις πιο ε, ε, αναπτυσσόμενες Τελειώνω, πρόεδρε. Τώρα πρέπει να δούμε τη διαφορά μεταξύ των ιδιωτικών κεφαλαίων και των hedge funds. Γιατί εκεί έχουμε καταρχήν μια ειδική συμπεριφορά των ε, κεφαλαίων κινδύνου. Εγώ θα ήθελα σε όλα τα κρατημέλη να έχουμε την ίδια, την ίδια νομοθεσία όπως σε εκείνες τις περιοχές που έχουμε το πιο δυναμικό κεφάλαιο κινδύνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Hans Peter Martin. Ναι, ευχαριστώ. Ε, θα εξοικονομήσω χρόνο. Γιατί πολλά ελέγξαν από του προλαλήσαντε. Εγώ έχω μόνο μία παράκληση προς τον εισηγητή. Αφήστε να εννοηθεί και το διαβάσαμε και στον τύπο πόσες επαφές υπήρξαν μαζί σας και προσπάθειες για επαχή επαφή. Θα μπορούσατε να μας πείτε πόσοι σας μίλησαν, σας έγραψαν και από αυτούς ποιο ποσοστό ε, έχουν την ε, έδρα των εταιριών τους στο Λονδίνο και πώς αυτό θα είχε επιπτώσει στις εργασίες σας, θα θέλετε να μας το πείτε. Δηλαδή, κατά πόσον λάβατε υπόψη επιχειρήματα που ακούσατε από έξω και σας έπεισαν. Κιάθριν Στάιλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον εισηγητή οι πληροφορίες σας ε, έδειξαν ότι πραγματικά αξίζει να σας εγκομιάσουμε για την πρότασή σας αυτή. Συμφωνώ με πολλά που είπαν οι προλαλήσατε συνάδελφοι. Εγώ θα συγκεντρώσω την προσοχή μου σε κάποια πιο προβληματικά θέματα. Αυτό το θέμα του short selling είναι κάπως αντιφατικά ε, διατυπωμένο. συνάδελφο Σάνι Μακάρθη εξετάζει το θέμα και θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια ε, μεταξύ της δικής της έκθεσης και αυτό. Όσον αφορά την συνέπεια με άλλα κείμενα και νομίζω ο κ. Κούτσος έθεσε το θέμα των ε, εταιριών επενδύσεων ε, συνδρήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Ο κύριος Κόντς αναφέρθηκε σε εξαιρέσει στις επενδυτικές αυτές εταιρείε. Ξέρω ότι το αναφέρεστε στο σημείο 16, 16 τρία συγγνώμη στην ε, συνέπεια με άλλα κείμενα θα πρέπει να φροντίσουμε ότι οι εταιρείε αυτές δεν είναι hedge funds ή ιδιωτικά κεφάλαια ότι θα πρέπει εδώ να έχουμε κάποια συνέπεια στην διατύπωσή μας και το θέμα του σεισμικού ε, κινδύνου που ό,τι υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια θα πρέπει νομίζω να μην το ε, διαγράψουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και προσβλέπω να συνεργαστούμε στους επόμενους μήνες. Πρώτα σε ευχαριστώ. Χάιλαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και ταυτόχρονα να ζητήσω συγγνώμη που επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο θα αναφερθώ μόνο στα αρνητικά ε, σημεία χωρίς να αγκομιάσω όλα τα θετικά που επέτυχε ο εισηγητής. Θα ήθελα να στιώσω την προσοχή μου στην αρχή της αναλογικότητας στην ε, νομοθεσία. Αυτό προσπαθούμε εδώ να ενδυναμώσουμε και η ενισχύα μου είναι ότι η εισηγητής αυτή τη στιγμή προτείνει να μην διατηρηθεί το κατόφλιο των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνω την σκέψη του, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αν αρχίσει κανένα να αναλύει τι θα σημαίνει αυτό, βλέπει ότι παραδείγματος για τη χώρα μου αυτό θα σημαίνει ότι ε, μια από ε, το κράτος ή ε, συστήματα συμμετοχής των εργαζομένων κλπ. κλπ. θα συμπεριληφθούν εδώ και αυτό δεν θα ήταν νομίζω πάρα πολύ αναλογικό γιατί ακριβώς προσπαθούμε να εξαφανίσουμε τον συστημικό κίνδυνο και όλα αυτά τα θέματα που σας προανέφερα δεν έχουν κανέναν ορατό συστημικό κίνδυνο και γι' αυτό είναι περιβολικό μου φαίνεται να τα περιλάβουμε εδώ. Ανησυχώ λοιπόν κάτι για την ιδέα να μην υπάρχει αυτό το κατόφλι στην οδηγία. Θα έπρεπε ίσως να το συζητήσουμε και να δούμε ποιε θα οι επιπτώσει για κάτι τέτοιο. Σε γενικέ γραμμέ, θα ήθελα να αναφέρω ότι το κείμενο βελτιώνεται, αλλά αυτό που εξακολουθεί να με ανησυχεί είναι ότι πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ελευθερήσουμε τον κίνδυνο και να μην τον εθαρρύνουμε. και δεν νομίζω ότι εδώ η οδηγία προβλέπει εκείνοι που έχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο ε, αντιμετωπίζονται πιο αυστηρά. Θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε και αυτό το θέμα της εμβέλειας της οδηγίας. Ευχαριστώ. σας ευχαριστώ κύριε Γεσέσκα. Όπω Όπως και άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να παρέμβω στο όνομα ενός ε, συναδέλφου που δεν είναι εδώ. Ε, ο συνάδελφος ε, μίλησε για την αναλογικότητα και υπάρχει μια δήλωση ε, που αφορά στην αναλογικότητα. Υπάρχει μια οδηγία που πρόκειται να εξετάσει το θέμα της αναλογικότητας. Ε, δεν ε, πρέπει να εξετάσουμε τις μεγάλες οντότητες που δεν συνεπάγονται συστημικούς κινδύνους 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν καταργήθηκε χωρίς να υποβληθεί μια εναλλακτική λύση, χωρίς να ληφθεί υπόψη, χωρίς να ληφθεί υπόψη, υπόψη μικρές επιχειρήσεις. Σας είπα λοιπόν ότι καταργήθηκε αυτή η πρόταση χωρίς να κατατεθεί εναλλακτική η οποία θα επέτρεπε να εξαιρεθούν ε, τα μικρά, τα επενδυτικά κεφάλαια μικρής εμβέλειας, κυρίως ε, τα ιδιωτικά. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό κινδυνεύουμε πάρα πολλά τα μικρά κεφάλαια θα πρέπει και αυτά να ληφθούν υπόψη. Έχουμε το άρθρο 11, το 12, το 13, το 16, το 17, 18, το 27 και στα επόμενα άρθρα δεν λαμβάνουν υπόψη, όπως σας είπα, τα μικρά κεφάλαια. Άλλο θέμα αφορά το άρθρο 14, οι προϋποθέσεις που θα διέπουν τα κεφάλαια. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά στα private equity ή στο καινοτόμο κεφάλαιο. Ε, δεν υπάρχει συστημικός κίνδυνος. Πάμε στο επόμενο θέμα που αφορά τις ε, τράπεζες ή τις οντότητες ε, παρακαταθήκων, των οποίων οι αρμοδιότητες διευρύνθηκαν σε σχέση με την αρχική πρόταση. Και βέβαια αυτές οι οντότητες δεν είναι καθοριστική σημασίας σε σχέση με τα ιδιωτικά κεφάλαια ή τα καινοτόμο κεφάλαια. Είναι επενδυτέ ε, μακράς πνοής, οι οποίοι δεν είναι εισηγμένοι. Και αυτοί δεν λαμβάνουν κερδοσκόπες αποφάσεις ε, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από τον ομιλητή να λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις τις οποίες μου ζήτησε να παρουσιάσω ο συνάδελφος που λείπει. Ο κύριος Πίτερ Σκίνερ, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ζαν Πολ, ο συνήθως ε, πάρα πολύ καλά εργαστήκατε, πολύ καλή η προσέγγισή σας. Βλέπω ότι στο τέλος όλοι σε ευχαριστούν. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αφαιρθώ στην προσέγγισή σου για την αναλογικότητα. Νομίζω, ε, το προσπάθησα και εγώ να το κάνω αυτό, να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ταμεία. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί να θέλει ένα ταμείο να είναι εκτός του πεδίου εφαρμογή του κανονισμού. Αυτή είναι μια πολύ καλή προσέγγιση. Και νομίζω ότι είναι πολύ ε, ε, οκνηρό το να βασίζεται κανείς ε, απλά σε κάποιους αριθμούς. Σωστά λοιπόν το θέτει. Το δεύτερο που θέλω να αναφερθώ είναι οι οντότητες παρακαταθήκων, τα αποθετήρια, τα depositories. Ε, ίσως αυτό το θέμα θα πρέπει να στηθεί σε κάποια άλλη οδηγία, αναφέρθηκε. Να, να πούμε όμως ότι όταν υπάρχουν ενδείξεις σε πρόκληση ζημιάς, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και εδώ ισχύει η εξή αρχή. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αφενός έχουμε τους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων και αφετέρου τις οντότητες παρακαταθήκων, που όμως σε ορισμένα κράτη-μέλη αυτά τα δύο είναι συνδεδεμένα. Οι επενδυτές παίρνουν τις αποφάσεις και αναλόγως ε, κάνουν λαμβάνουν, κάνουν κάποιες επενδύσεις και οι αρμόδιοι για την ε, εναπόθεση, αυτοί έχουν και αυτοί τις δικές τους επενδύσεις, δικές πληροφορίες. Όταν μιλάμε για ένα δις ε, δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στα, στις οντότητες παρακαταθήκων και ε, στους ε, επενδυτές. Πρέπει να τα διαχωρίσουμε. Αυτό είναι προς όφελος του επενδυτή. Δεν μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε αργότερα να εκπονηθεί μια οδηγία. Ήδη έχουμε πάρα πολλούς ε, επενδυτές που πολλούν άμεσα. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους επενδυτές ε, από ε, επικίνδυνα πράγματα ή Λέμαν παραδείγματος χάρη. Χάθηκαν δισεκατομμύρια γιατί δεν ε, μπορέσαμε να αποδείξουμε ότι υπήρχε ολιγορία και εκ μέρους των επενδυτών αλλά και εκ μέρους των αποθετηρίων. Είναι λοιπόν σημαντικό να προστατεύσουμε τους επενδυτές ε, των ε, ε, παρακαταθήκων από αυτούς που επενδύουν επικίνδυνα κεφάλαια. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Γάλλοι που ενεπλάκησαν στην υπόθεση Μέντοφ, γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό για μας Ευρωπαίους να μην ξαναβυθιστούμε. Η Αιλίν έχει το λόγο. Συγγνώμη, λάθος, κύριε Γουότμαν Κόλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι σύντομη, ε, κυρίως στις ευχαριστίες μου, όμως ε, τελικά το να μην πλατιάζει κανείς ευχαριστίες, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ευχαριστεί, εκ βάθους. Θα εστιάσω την προσοχή μου στα σημαντικά. Ε, να δούμε κατά πόσον η έκθεση ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Εγώ προσωπικά πιστεύω, όπως και ο εισηγητής, το πεδίο εφαρμογής να παραμείνει αυτό που προτείνει. Πρόκειται και για κάποια άλλα θέματα. Στην Ολλανδία, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν συνταξιοδοτικά ταμεία τα οποία έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες, κατ' ουσίαν όμως πρόκειται για ένα και μόνο συνταξιωτικό ταμείο και δεν θέλουμε να εμπίπτουν εκεί τα πάντα. Είπατε ότι πρέπει να καταργηθεί το κατώτατο όριο, το κατόφλι. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κατά πόσον αυτό είναι λογικό. Δηλαδή, κατά πόσον πράττοντας κάτι τέτοιο, υπάρχει ενδεχομένως ο κίνδυνος να υπονομεύσουμε τον κανονισμό. Εγώ δεν πιστεύω ότι μεγάλα επενδυτικά ταμεία θα διασπαστούν για αυτό το λόγο σε μικρότερα, επειδή τα μικρότερα υποτίθεται ότι δεν ελέγχονται. Δεν έχω σαφή εικόνα για το τι ακριβώς ε, συμβαίνει με αυτή την περίφημη αναλογικότητα. Κατ' ουσίαν, πρόκειται για το εξής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποκλείσουμε τον δεχόμενο κινδύνων και να προσφέρουμε ως το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια. Όσον αφορά λοιπόν την αναλογικότητα. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά για να έχουμε μία πραγματική διαφοροποίηση ανάμεσα στα πραγματικά επικίνδυνα αμοιβαία κεφάλαια και τα υπόλοιπα. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να περιορίσουμε ως δυνατόν το διοικητικό άχθος. Τελευταία μου παρατήρηση. Πρόκειται για τις ε, τρίτες χώρες. Έχω να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, είναι αλήθεια σωστό να λέμε τα μία από τρίτες χώρες δεν μπορούν να αποκτήσουν το ευρωπαϊκό διαβατήριο. Βεβαίως και πρέπει να διεξάγονται οι έλεγχοι, αλλά απλά το να κλείσουμε την πόρτα, αυτό για μένα προχωράει πάρα πολύ. Κατόπιν όσον αφορά τις ε, ιδιωτικές επενδύσεις, private placement, Εκεί το κράτος μέλος δύναται να συνάψει διμερείς συμφωνίες. Μερικοί αυτό ενδεχομένως να το βλέπουν θετικά. Αλλά για σκεφτείτε τι θα συμβεί, τελικά θα προκύψει ανταγωνισμός ανάμεσα στα ίδια τα κράτη-μέλη. Είναι προφανές ότι τα ταμεία θα μεταφερθούν στο Λονδίνο και τι φαντάζεστε, θέλουμε πραγματικά να υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Μήπως λοιπόν θα ήταν λογικό να αναζητήσουμε κάποια λύση και για τα ταμεία των τρίτων χωρών. Δεν έχω να προτείνω κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να αναζητήσουμε μια τέτοια λύση. Νομίζω ότι ελέγχθησαν τα περισσότερα και σωστή προσέγγιση του κυρίου ε, Γκοζέ... για να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Μάρτιν. Κοιτάξτε, νομίζω ότι συναντήθηκε με όλους τους διαχειριστές αμοιβαίων από όλα τα, ε, τις ε, σημαντικές μητροπόλεις αγοραπολισιών. Αυτό που βρίσκω σημαντικό είναι ότι συναντήθηκε και με επενδυτέ από το Λονδίνο. Ίσως λοιπόν μπορούμε να θέσουμε τέλος σε αυτή τη θεωρία περί σκευωρίας ότι προσπαθούμε να εξαφανίσουμε το Λονδίνο. Δεν συμβαίνει αυτό. Και ο κ. Μπαρνιέ έχει αναγνωρίσει τη σημασία του Λονδίνου και τη σημασία όλων των επενδυτικών κέντρων. Πρέπει να μάθουμε το μάθημά μας από την κρίση, να μπορούμε να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το ότι ο εισηγητής ε, μιλάει για μια ζωντανή καινοτόμο προσέγγιση, ένα καινοτόμο τομέα. Είναι καλό που μιλάμε για την αναλογικότητα. Με αυτή την προσέγγιση νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε κάποιες επιλογές και επιλογή είναι ε, αυτό που έχει υποθεί επανειλημμένα ότι δεν υπάρχει συστημικός ε, κίνδυνος ε, με αυτά τα κεφάλαια. Αλλά τι θα κάνουμε, θα τα Ξερέσουμε από την νομοθεσία. Θα είμαστε μήπως αναλογικοί ή αυτό που είπε ο κύριος Χουκμαρκ ότι θα πρέπει ενδεχομένως να αναζητήσουμε ένα διαφορετικό καθεστώς ε, διαφάνειας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Καλύτερα να το λύσουμε έτσι από γραφειοκρατικού κανόνε, οι οποίοι κάποια στιγμή θα εξοντώσουν αυτά τα επενδυτικά ταμεία και θα υπονομεύσουν τη ζωντάνια τη Ευρώπη, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Για τι τρίτε χώρε, Χαιρετίζω το γεγονό που λέει ο κύριο Γκοζέ ότι θα πρέπει οι επενδυτέ να έχουν την ευκαιρία και την ελευθερία να επενδύσουν και σε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει μία ε, συμφωνία για την ανταλλαγή πληροφοριών, είτε θα πρέπει να ελέγχονται αυτές οι επενδύσεις. Υπάρχουν βέβαια πρακτικές ε, δυσκολίες, αναφέρθηκαν μερικές εξ αυτών. Το ερώτημα που έχω εγώ είναι περισσότερο ένα ερώτημα για πληροφόρηση, γιατί ξέρω την απάντηση. Τι θα γίνει με αυτά τα ταμεία των τρίτων χωρών που επενδύουν ότι το αποθετήριο θα πρέπει να βρίσκεται στη χώρα από την οποία ξεκινούν οι επενδύσεις. Δεν νομίζω ότι ε, είναι ρεαλιστικό να πιστεύει κανείς ότι οι τρίτες χώρες θα δεχθούν να μεταφέρουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι καλό να έχουμε συγκεντρωτισμό των αποθετηρίων. Ε, ίσως από εκεί να προκύψει μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά, αλλά σε επίπεδο αρχή, πραγματικά εκτιμώ τη δουλειά που έκανε ο Ζαν Πολ. Είναι πολύ καλή δουλειά του, ισόρροπη και είναι ανοιχτή στο ε, να βρούμε την λύση που όπω λέει και ο ίδιο να είναι η εξισορρόπηση των συμφερόντων να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί για να αναστείλουμε οποιοδήποτε συστημικό κίνδυνο υπάρχει σε αυτόν τον τομέα. Πολύ ωραία. Ε, κανείς άλλος δεν θα λάβει το λόγο. ελέχθησαν τα περισσότερα και εγώ θα ήθελα απλά και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι ένα πολύ καλό βήμα προς τα εμπρός. Ε, όπως και άλλοι ανέφεραν θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε ορισμένους ε, τομείς ε, στα ιδιωτικά επιχειρηματικά κεφάλαια, στα καινοτόμα επενδυτικά κεφάλαια και σε πάρα πολλά άλλα. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω την ε, Κομισιόν τώρα να μας δώσει μία απάντηση και κατόπιν ο Ζαν Πολ θα μπορέσει να ανακεφαλαιώσει. Ε, δεν θα πρέπει όμως ή δυνατόν να μιλήσετε πάνω από τέσσερα λεπτά σας παρακαλώ πολύ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι. Θα προσπαθήσω να μιλήσω και λιγότερο από τέσσερα λεπτά. Γιατί θα ήθελα απλώ να χαιρετήσω την έκθεση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Η Κομισιόν παρανοχή στην έκθεση του κ. Κόζε και τη συνεργασία που η Ελλάδα χώρα με τον ίδιο και με άλλα μέλη εδώ της, του σώματο. Η έκθεση μου φαίνεται ότι το γενικό κανόνα κινείται προς την κατή, σωστή κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση της Κομισιόν δηλαδή. Όλο που βέβαια υπάρχουν και διαφορές. για ορισμένες πτυχές και μερικές ε, αποκλήσεις βέβαια που υπάρχουν αλλά πιστεύω ότι η συζήτηση που έγινε μέχρι στιγμής και που ήταν πάρα πολύ επικοδομητική θα συνεχίσει και θα μας επιτρέψει να εξαλείψουμε τις διαφορές. Θα ήθελα καταρχήν να τονίσω τις συγκλήσεις, είναι σημαντικές, γιατί αναφέρονται σε στοιχεία πολύ σημαντικά, όπως πρέπει την υποστήριξη στην ύπαρξη νομοθεσίας, στην ανάγκη δηλαδή διακανονισμού του τομέα, που δεν ήταν ε, ένα κεκτημένο στοιχείο της συζήτηση πριν από μερικούς μήνες. Κατόπιν, προφανώς οι στόχοι. Οι στόχοι μας φαίνονται ότι το συμμεριζόμαστε από καινού. Οι κύριοι στόχοι, οι τρεις κύριοι στόχοι της θέσης της Κομισιόν φαίνεται ότι οθετούνται από τον κύριο Κοζέ στην έκθεσή του. Ιδίω στον έλεγχο του συστημικού κινδύνου, την προτεστασία του καταναλωτή και επίσης η πτυχή της εσωτερικής αγορά. Αναφέρεται κυρίω στην υποστήριξη τη ιδέας για ένα διαβατήριο ευρωπαϊκό. δύο εφαρμογέ. Ξέρετε και το είπα ήδη. Αυτό που λέγεται All Encompassing Approach ήταν ένα βασικό στοιχείο της ε, πρότασης που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την εξαντλησμό του διχειριστή. Κατόπιν έχουμε εδώ λειτουργικό τομέα που μας φαίνεται ότι παρουσιάζεται σωστά στην ε, έκθεση όσον αφορά τις απαιτήσεις που υπάρχουν για τον ζεβασμό των όριων, για τους ίδιους πόρους. Πολλά δηλαδή, πολλά στοιχεία που μας ενδιαφέρουν. Υπάρχουν θέσεις του κυρίου Ζωρές, ε, χαιρόμαστε γι' αυτό. Υπάρχουν και διαφορές ε, δεν μπορώ να τι αναπτύξω όλα για να σεβαστώ τα τέσσερα λεπτά. Θα ήθελα απλώ να τονίσω ένα σημείο το οποίο ίσω σα εκπλήξει, και το οποίο ακόμα πρέπει μπορεί να λύγουν. Πρόκειται για το θέμα των τρίτων χωρών, που πολλοί από του παρεμβαίνοντε θεωρούνται σαν ένα σημαντικό ε, σημείο σε μια κύρια δυσκολία του φακέλου. Ε, η ιδέα των να αφαιθούν τα πράγματα στην αρμοδιότητα των κρατών μελών είναι μια προκλητική ιδέα και πολύ ρεαλιστική. Αλλά δεν θεωρούμε ότι αυτή είναι μια πρόταση που δεν έχει κανένα κίνδυνο του αντίον. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Να μείνει δηλαδή η επιλογή η Ευρώπη να γίνει φρούριο ή σουρωτήρι, να παραμείνει στην ε, διακριτική ευχαίρεια κάθε κράτους μέλους, με αποτέλεσματα απρόβλεπτα όσον αφορά το ε, επίπεδο πεδίο παιδής, ε, Λοιπόν, σας ευχαριστώ για αυτά που έχετε κάνει μέχρι στιγμής και σας καλώ όλους να σκεφτείτε το θέμα του. Σταματώ εδώ, 3 και 57 λεπτά μίλησα. ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Ο εισηγητής έχει το λόγο αν θέλει να πει κάτι. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Σύμφωνα με τη μέθοδο μου, δεν θέλω να προασπίσω την έκθεσή μου, θα κάνω μερικά σχόλια μόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπο πυρογνώμονε και συνεργάτε τη γραμματεία που με βοήθησαν στην προετοιμασία τη έκθεση αυτή. Κατόπιν θα ήθελα να καθησυχάσω τον κύριο Μάρτιν, ο οποίο προφανώ ανησυχεί για την υγεία μου και α, με ρωτάει μήπω υποδέχτηκα πολλού, Εγώ όσου μου το ζητάει τον δέχομαι. Για αυτή την έκθεση πολλοί ήταν. Πού ήταν αλλά και στι περασμένε έκθεσει ήταν πολλοί. Γιατί νομίζω ότι η συμβολή εκείνο που έρχονται να μας μιλήσουν είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρουμε ποιον, ποιον εκπροσωπούν, ξέρουμε ποια είναι τα συμφέροντά τους και είναι χρήσιμο να τους ακούσουμε. Γιατί ακούγοντας διαφορετικά συμφέροντα μπορεί κανένας να δημιουργήσει μια άποψη.